So, good afternoon everybody and welcome back. Καλώς ήρθατε και πάλι. Καλησπέρα σας. Αυτή είναι η πρώτη μας ε, συνεδρίαση μετά από τις ε, διακοπές των Χριστουγέννων. Καλώς ορίσατε λοιπόν και πάλι στην Επιτροπή Αναφορών και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ελπίζουμε ότι η νέα χρονιά δεν είναι καρποφόρος και μια καλή χρονιά. Έχουμε ακόμη τέσσερις συνεδριάσεις στην Επιτροπή μας πριν ε, να διαλυθεί το Κοινοβούλιο και πριν την ε, προεκλογική εκστρατεία και ίσως ε, κάποιοι να ξανάρθουμε μετά τις εκλογές. Αλλά όπως και να έχει όλοι θα κερδίσουν γιατί και όσοι δεν επενεκλεγούν θα κερδίσουν την ελευθερία τους. Όλοι είμαστε ε, νικητές, θα κερδίσουμε μια νέα έδρα, θα κερδίσουμε την ελευθερία μας. Λοιπόν, να επικεντρωθούμε τώρα σε όσα έχουμε να συζητήσουμε σήμερα. Είναι βεβαρημένη η ημερήσια διάταξη. Καταρχήν, να περάσουμε στην ημερήσια διάταξη και να δούμε τι υπάρχει εδώ. Έχουμε δύο αιτήματα τροποποίησεων, τροποποίηση συγγνώμη, της ημερήσιας διάταξης, να αναβληθεί το σημείο 21. Κατόπιν αιτήματο ε, του αναφέροντα γιατί δεν μπορεί να παρευρεθεί τον Ιανουάριο και επίση αναβολή του σημείου 27 κατόπιν αιτήματος της ΓΚΟΕ. Μπορούμε να το πράξουμε αυτό, να αναβάλουμε τα δύο αυτά σημεία. Σας ευχαριστώ πολύ. Όχι, Πίτερ. Ε, δεν θα θέλαμε να αναβληθεί το υπαριθμό 27. Είμαστε λοιπόν αντίθετοι με την αναβολή. 27 έτσι δεν είναι. 27. 21 λέτε. Με συγχωρείτε για τη σύγχυση. Είμαστε κατά της αναβολής της αναφοράς που περιλαμβάνεται στο 21. Ε, λοιπόν, εκεί είμαστε αντίθετοι. Να παραμείνει στην ημερησία διάταξη θέλουμε. Άρα θα θέλατε να διατηρηθεί το 21. Αλλά θα θέλατε να αναβληθεί το 27. Αυτό μου λέτε ή θέλετε να αναβληθούν και τα δύο. Θέλετε να αναβληθεί το 21. Θέλετε να παραμείνει. Να παραμείνει, ναι. Ωραία. Το 21 κανείς δεν έχει ζητήσει να αναβληθεί. Ο αναφερόμενος δήλωσε ότι δεν μπορεί να προσέλθει σήμερα. Πρέπει λοιπόν να ψηφιστεί για να υπάρξει σαφήνεια. Ποιο θα ήθελε να συμφωνήσει να αναβληθεί το 21, γιατί ο αναφερόμενος δεν μπορεί να είναι παρόν. Η πράσινη και η FTD ποιο θέλει να συζητηθεί ακόμη και εάν είναι απόν ο αναφερόμενος, το Λαϊκό Κόμμα. Ας ε, μετρήσουμε τις ψήφους. Οι σοσιαλιστές δεν ψηφίζετε, έτσι δεν είναι. Επαναλαμβάνω, επαναλαμβάνω γιατί φαίνεται πως δεν είναι σαφές. Ποιος θα ήθελε να αναβληθεί το 21. Σοσιαλδημοκράτες, Γκουε, Πράσινη και η FTD. Ποιος θέλει να διατηρηθεί το υπαριθμό 21, ακόμη και αν ο αναφερόμενος δεν είναι παρόν το Λαϊκό Κόμμα. Κάντε παρακαλώ τον υπολογισμό. You know what? I need to bring it to an... Νομίζω ότι χρειάζεται να γίνει ηλεκτρονικά η ψηφοφορία για να είμαστε και πιο σίγουροι. Okay. So. Η πρόεδρος πάλι. Σας παρακαλώ. Εάν ψηφίσετε ναι, σημαίνει αναβολή. Αν ψηφίσετε όχι, δηλαδή το κόκκινο κουμπάκι, τότε θα παραμείνει σήμερα στην ημερήσια διάταξη. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ε, εννοώ βέβαια την ημερήσια διάταξη αύριο. Αρχίζει λοιπόν η ψηφοφορία. Ωραία. Δέκα λοιπόν να αναβληθεί 8 κατά της αναβολής. Άρα αναβάλλεται το 21. Τώρα, 27. Να κάνουμε το ίδιο. Τώρα στην περίπτωση αυτή, το 27 έχει ζητήσει η Γκουε να αναβληθεί. Όσοι λοιπόν είναι υπέρ της αναβολής, να πατήσετε το πράσινο κουμπί και όσοι θέλετε να παραμείνει στην ημερήσια διάταξη να πατήσετε το κόκκινο κουμπί. Αν είστε υπέρ της αναβολής, πράσινο. Αν θέλετε να μείνει στην ημερήσια διάταξη, κόκκινο. Α, μάλιστα. Ισοψηφία, διότι ε, είναι ισοψηφία, άρα απορρίπτεται. Άρα παραμένει στην ημερήσια διάταξη. Καλώς. Έτσι λοιπόν θα κάνουμε. Τώρα, αν δεν έχετε άλλε ενστάσεις ε, να ε, υποβάλλετε, ας εγκρίνουμε την μέση διάταξη με τις αλλαγέ που έχετε επιφέρει. Τώρα, τα πρακτικά της 27 η Νοεμβρίου έχουν διαβιβαστεί, έχουν διαβαστεί, δεν βλέπω να υπάρχουν ενστάσεις, τα εγκρίνετε λοιπόν, ωραία. Δεν έχω ανακοινώσεις να κάνω, θα τις κάνω αύριο το πρωί. Επίσης δεν έχουν ζητηθεί διάφορα. Άρα, προχωρώ αμέσως στην, στην, στην ψηφοφορία. Ψηφοφορία. Για την εφαρμογή του χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αφού ήδη έχετε βάλει τις κάρτες σας, εύκολο είναι να ψηφίσετε αμέσως. Τροπολογία 1 υπέρ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 αποχές απορρίπτεται 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 9 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 11 υπέρ Θέλετε επαλήθευση για την 10 τροπολογία 10 Αρχίζει η επαλήθευση τώρα λοιπόν, η ηλεκτρονική επαλήθευση. Αρχίζει τώρα. Τέλος. Εγκρίνεται. Η 11 τώρα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 12 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μια στιγμή 18 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 25 σε δύο τμήματα. Πρώτο υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 28 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 30 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, συμβαστική 6 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 32 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 33 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 34 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 35, αν με συγχωρείτε αυτό εκπίπτει, συμβαστική 7 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 44 υπέρ κατά αποχές δεν φαίνεται καλά από τα χέρια. Χρειάζεται λοιπόν ηλεκτρονική επαλήθευση 44. Τέλος εγκρίνεται. Από τώρα παρακαλώ ψηλά τα χέρια. 45 υπέρ. Κατά. Αποχές. Και εδώ χρειάζεται επαλήθευση. Για να δούμε. Εγκρίνεται. Απέχει το Λαϊκό Κόμμα. Η προφορική τροπολογία 47 δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 48 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 50 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 51 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 52 εκπίπτει 53 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 54 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 55 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 59 υπέρ κατά αποχές δεν μπορώ να δω καθαρά νομίζω ότι απορρίπτεται 60 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 65 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 64 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 66 θέλετε επαλήθευση για την 64. Ας κάνουμε λοιπόν επαλήθευση με ηλεκτρονική ψηφοφορία. 64. Τέλος. Εγκρίνεται έστω και με μία ψήφο διαφορά. Η 66 εκπίπτει διότι εγκρίθηκε 64. 67 υπέρ. 67 λέω υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 68 εκπίπτει 69 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 70 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 71 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 72 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 73 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 74 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 76 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 78 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 79 α, α μια στιγμή 78 ηλεκτρονική ψηφοφορία επαλήθευσης. Τέλος, απερίφθη 79 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και η τελική ψηφοφορία τώρα για το σχέδιο γνωμοδότησης, όπως τροποποιήθηκε, ηλεκτρονικά, αρχίζει η ψηφοφορία, ξαναλέω είναι η τελική ψηφοφορία, Τέλος. Εγκρίνεται. Χωρίς πολύ μεγάλη διαφορά βέβαια. Now, uh, those... Τώρα, Όσοι από εσά ε, θα θέλατε να αποχωρήσετε, να πάτε σε άλλη αίθουσα ή να πιείτε ένα καφέ, παρακαλώ να το κάνετε με ήσυχο τρόπο, ώστε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε με την αναφορά. Έχετε λίγα ε, λεπτά στη διάθεσή σας για να μπορέσετε να βγείτε από την αίθουσα. coming. Okay, the petitioner is not here. No, no, exactly. Exactly, exactly. Now, dear friends. Αγαπητοί φίλοι, ας προχωρήσουμε. Στην αναφορά 0207 για την ε, μόλυνση της παραλίας ε, Whitburn στο Ηνωμένο Βασίλειο. Για λόγους υγείας δεν μπορεί να παρευρίσκεται ο αναφέρον. Του στέλνουμε τις καλύτερες ευχές μας διαπηρεαστικά και θα ζητήσουμε από τη συνάδελφο την Κίτεν Ντάρλινγκ να διαβάσει την δήλωση του αναφέροντος ε, μέσω της δική τη φωνής θα ακούσουμε τον αναφέροντα για πέντε λεπτά έχει το λόγο Ευχαριστώ Πρόεδρε όπως είπατε, δυστυχώς ε, ο κύριος Μπομπλάτιμερ δεν μπορεί να βρίσκεται εδώ σήμερα ε, γιατί πέστη μια εγχείρηση και δεν ε, έχει πλήρη κινητικότητα. Έτσι λοιπόν του στέλνουμε και εμείς ευχές για περαστικά. Είναι μια υπόθεση που τρέχει εδώ και καιρό. Το αρχική καταγγελία στην Κομισιόν ήταν το 2000. Είχαμε απόφαση από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο το 2012 και ε, εν τέλει αφορά την ικανότητα του συστήματος ε, ε, ε στην δική μου ε, περιφέρεια, εκλογική περιφέρεια και τον ε, αντίκτυπο που έχει στην ρήπανση των θαλασσών. Νομίζω ότι δεν σου αξίζει να υπάρχει τέτοιο θόρυβο στην αίθουσα. Όσοι δεν θέλουν ε, να βρίσκονται εδώ, να αποχωρήσουν τώρα, παρακαλώ. Μπορείτε να συζητήσετε εκτός της αιθούσης, παρακαλώ, για να μπορέσουμε κι εμείς να συνεχίσουμε όπως πρέπει με την εξέταση της αναφοράς. And there is a large group of visitors coming. Και έχουμε και μια μεγάλη ομάδα επισκεπτών. Δεν ξέρω ποιοι είστε ή από πού έρχεστε, αλλά καλώ ήρθατε στην ε, συνεδρία τη Επιτροπή μα. So, Jude, I think that there is now. Jude, νομίζω ότι τώρα μπορεί να πάρει το λόγο. Θα διαβάσω λοιπόν ακριβώς ε, αυτά που μου ζήτησε να διαβάσω αναφέρον στην Επιτροπή αποτελεί απάντηση στην απάντηση της Κομισιόν της 31 Οκτωβρίου 2018. Η Κομισιόν ε, βασίζεται σε πληροφορίες ε, που ε, έλαβε από την Authority Water Limited και έχουμε 298.000 σε 8 μήνες το 2018. Αυτά τα δεδομένα ε, πρέπει να τα αμφισβητήσουμε. Δηλώνεται ότι τέτοιες απορρίψεις ε, προέκυψαν από ισχυρή ε, βροχή χιονόπτωση, αλλά δεν υπάρχουν αποδείξεις. Το 2018 ήταν μία από τις πιο ξηρές χρονιές, τουλάχιστον 10% κατά μέσο όρο στην περιοχή μας και η χιονόπτωση ήταν μόνο 6 με 10 εκατοστά σε 5 μέρες. Φαίνεται ότι ο σκοπός του συστήματος του Whitman ήταν απλώς να σεβαστεί την οδηγία ε, χωρίς να υπάρχουν απορρίψεις στη θάλασσα. Έχουμε δύο σημαντικές αλλαγές στην καταγραφή των δεδομένων και σημαίνει ότι δεν μπορούμε να πιστέψουμε τις πληροφορίες που δόθηκαν στην Κομισιόν. Ισχυρίζονται καταρχήν ότι ε, στη μελέτη του 2010 για την Whitburn Steel LSO έχουμε ε, απορρίψεις για λιγότερο από 30 λεπτά και θεωρούνται αυτές όσο μη απόρριψη. Όμως, αν έχουμε μία απόρριψη 25 5 λεπτών θα είχαμε 4.500 ε, κεμικά μέτρα, 4.500 ε, τόνους ε, λιμάτων που δεν καταγράφονται. Δεύτερον, έχουμε τη διατύπωση της απάντησης του Ηνωμένου Βασιλείου στην αιτιολογημένη γνώμη της Κομισιόν που λέει αν προβλέπετε βροχή, η Northumbrian Water Limited θα διάσει τη δεξαμενή στα 2.000 κυβικά μέτρα. Η δεξαμενή περιλαμβάνει 7.000 κυβικά μέτρα πριν να υπάρξει αυτόματη, αυτόματο άδειασμα, δηλαδή αυτό σημαίνει ότι 4.500 κυβικά μέτρα μπορούν να απορριφθούν σε λιγότερο από 30 λεπτά. Έτσι λοιπόν και πάλι δεν θα καταγραφούν. Η δική μας εμπειρία είναι ότι έχουμε πολύ περισσότερες απορρίψεις από αυτές που καταγράφονται και η συνέπεια είναι η συνεχής ε, παρουσία ε, λιμάτων υπονόμων στην παραλία και στα παράκτια ύδατα. Ε, τα έργα αποκατάσταση, όπω ζητήθηκαν από το δικαστήριο, ήταν ελάχιστα και ήταν ε, τα εξή. Χτίστηκε ένα φράγμα από τούβλα προκειμένου να μπορέσει να κρατήσει πίσω τι ροέ στο βασικό υπόνομο. Δήλωνε η απόφαση ότι θα έπρεπε να αυξηθεί η ικανότητα του υπονόμου, όμω αυτό δεν έγινε. Υπήρξε επιπρόσθετη δεξαμενή ε, αποθήκευσης που, που συνδέθηκε με το σύστημα υπονόμων, αλλά όχι για τις καταιγίδε. Επίσης, ε, αντλίες ε, πολιτοποίησης τοποθετήθηκαν στα αντιλιοστάσια. Παρόλα αυτά έχουμε πλαστικά υγειονομικά τεμάχια που περνάνε μέσα και αποκαλύπτουν ότι υπάρχουν απόβλητα στην παραλία. Επίσης, ε, πολλές από τις πληροφορίες που χρησιμοποιήθηκαν ε, δεν ήταν σωστές. Αυτό οδήγησε σε μη κατάλληλες βελτιώσεις σε ένα κατάλληλο σύστημα που δεν μπορεί να επεξεργαστεί τα λύματα από ένα αυξανόμενο πληθυσμό και επομένως υπάρχουν απορρίψεις απευθείας στη θάλασσα. Αν και η Κομισιόν δεν ε, έχει ερευνητικές αρμοδιότητες, δεν μπορεί απλώς να εξαρτάται σε δεδομένα που δίνει ο παραβάτης, αλλά θα πρέπει να ζητήσει ανεξάρτητα στοιχεία, διαφορετικά η οδηγία για την επεξεργασία των αστικών λιμάτων είναι ανοιχτή στην ερμηνεία και άχρηστη. Ε, αν ε, η Κομισιόν ε, είχε προσβάλει τα στοιχεία αυτά στο δικαστήριο, δεν θα παρουσίαζα σήμερα αυτά τα στοιχεία στη δική σας Επιτροπή. Τέλος, τώρα είναι επιτακτικό μία πλήρης και ανεξάρτητη επισκόπηση της δομής του συστήματος των υπονομών υλοποιηθεί ε, για να διασφαλίσει όχι μόνο ότι είναι κατάλληλο το σύστημα για εξυπηρετήσει το σκοπό, αλλά και ότι έχει και την ε, ικανότητα για τα 5.000 ακόμα σπίτια όπω προτείνεται. Δεν είναι αλήθεια όπω δηλώνει η Κομισιόν ότι αυτό αφορά μόνο ε, την εθνική νομοθεσία. Έχουμε απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και απέτησε να υπάρξει βελτίωση στην απόφαση. Τώρα δεν υπάρχουν τέτοιες βελτιώσεις και το σύστημα συνεχίζει να παραβιάζει την οδηγία για την επεξεργασία λιμάτων, καθώς το σύστημα Σάντερλαντ δεν ε, ε, επεξεργάζεται όλες τις ροές. Αυτά θα είχε πει ο αναφέρον, αν μπορούσε να είναι εδώ σήμερα το απόγευμα. Ευχαριστώ, Τζούντ. Είναι μία από αυτές τις υποθέσεις που σκέφτομαι αυτή θα είναι η τελευταία υπόθεση που θα, θα μας απασχολήσει με το σωστό τρόπο πριν φύγει το Ηνωμένο Βασίλειο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σίγουρα το δικαίωμα στην αναφορά είναι ένα από αυτά τα δικαιώματα που έχουν όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες και χαίρομαι που ο Ρόμπερτ Λάτιμερ χρησιμοποίησε αυτό το δικαίωμα και υπέβαλε αναφορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τώρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κυρία Γκρός, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει το λόγο. Σας ακούμε. Λάβαμε κι εμείς ένα αντίγραφο της δήλωσης του κυρίου Λάτιμερ ε, που διαβάσατε. Δεν διαφωνούμε με τα όσα λέει ο κύριος Λάτιμερ. Δηλαδή, οι βελτιώσεις που έγιναν, τα έργα που έγιναν, δεν βελτίωσαν επαρκώς ε, ε, το σύστημα ε, όπως ελπίζαμε και ελπίζε και ο αναφέρον. Είχαμε κάποια συζητήσει με τον Δωμένο Βασίλειο. Δεν συμφώνησε 100% σε ό,τι αφορά τις βελτιώσεις αυτές που χρειαζόταν στην περιοχή του Whitburn. Μετά από κάποιες συζητήσεις συμφώνησαν να κάνουν ουσιαστικές επενδύσεις για να βελτιώσουν το σύστημα υποδοχής λιμάτων είναι μια πρωτότυπη, πρότυπη υπόθεση που έφερε η Κομισιόν αυτή στο δικαστήριο. Ε, λάβαμε πολλές αναφορές, όχι μόνο του, αυτή του κυρίου Λάτιμερ για το Whitburn, αλλά και για άλλες περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου και συνειδητοποίησαμε ότι παρότι το Ηνωμένο Βασίλειο έφτιαξε εγκαταστάσεις επεξεργασίας λιμάτων ε, των ε, αποχε... αποχετεύσεων, δυστυχώς υπάρχει υπερχείληση ανεπεξέργαστων, ακατέργαστων κλιμάτων σε μεγάλο βαθμό. Το Whitburn ε, αντιμετωπίζει το πρόβλημα που παρουσίασε ο κύριος Λάτιμερ. Περιμέναμε μέχρι να γίνουν όλα αυτά τα βελτιωτικά έργα. Ε, ολοκληρώθηκαν στο τέλος του 2018 για να δούμε αν αυτές οι ε, βελτιώσεις ήταν αποτελεσματικές. Έπρεπε να περιμένουμε τα δεδομένα των διαρροών, τα οποία α, παρουσίασε ο κύριος Γουί. Ε, εδώ στην Επιτροπή Αναφορών από τον κύριο Λάτιμα. Και υπάρχουν προβλήματα παρά τις βελτιώσεις. Ε, οι βελτιώσεις δεν είναι ένας απλός ε, τείχος. Ε, αυξημένη δυνατότητα αποθήκευσης υπάρχει. Ε, επίσης, ε, κάποιες ε, περιοχές εκ των υστέρων απομονώθηκαν, ας πούμε, από, το, από τους υπονόμους αλλά παρόλα αυτά οι βελτιώσεις δεν ήταν τόσο σημαντικές, ε, τόσο πλήρε όσο ελπίζαμε. Στην επόμενη φάση θα πρέπει να δούμε ε, εάν η Επιτροπή θα προχωρήσει με περαιτέρω διαδικασία επιπαραβάση. Είναι υποσυζήτηση το θέμα. Σας ευχαριστώ για τη σαφέστατη δήλωση. Περαιτέρω διαδικασία επιπαραβάση προβλέπετε, προβλέπεται, δηλαδή θα συνεχίσει η υπόθεση. Τώρα θα δώσω το λόγο στους βουλευτές. Η Θέλει να ξαναμιλήσει. Όχι εκπροσωπώντα τον κύριο Λάτιμερ. Λοιπόν, ζητώ συγγνώμη που ξαναπέραν το λόγο. Θέλω να πω τις δικέ μου απόψει τώρα. Καλωσορίζω τη δήλωση της Κομισιόν. Ήταν μια δύσκολη και μακρά υπόθεση αυτή για όλους όσους συμμετείχαν και μία από τις πιο βρώμικες ε, των βρώμικων ε, περιοχών της Ευρώπης. Εμείς στα βόρειο-ανατολικά, από μια άθλια κατάσταση σε ό,τι αφορά την ποιότητα του νερού, φτάσαμε σε μια εκπληκτική κατάσταση σε ό,τι αφορά την φυσική μας ομορφιά, ε, χάρη στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Ε, η περιβαλλοντική νομοθεσία ε, της Ευρωπαϊκή Ένωση, ειδικά η νομοθεσία για το νερό, ήταν σημαντική για να βελτιώσουμε τους ποταμούς, τις παραλίες και το σύστημα ίδρευσης και να κάνουμε περισσότερες επενδύσεις ε, στην επεξεργασία των αστικών λιμάτων. θα πρέπει να επαγρυπνούμε, ούτω ώστε να μην υπαναχωρήσουμε και οι δεσμεύσεις που έχουν αναλυφθεί από την ΕΒ ως κράτος μέλος να εφαρμοστούν όπως πρέπει. Θέλω να αποτίσω φόρο τιμής στον Bob Λάτιμερ και σε όλους όσους ε, συμμετείχαν σε αυτές τις εκστρατείες ε, που έκαναν πραγματικότητα την ευρωπαϊκή ε, περιβαλλοντική νομοθεσία. Γιατί πρέπει να είσαι πραγματικά πεισματωμένος, να επι, επίμονος, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά συμφέροντα. Αν σε ενδιαφέρει όμως η κοινότητά σου, η περιοχή που μένεις και αντιμετωπίζεις τέτοιες υποθέσεις που είναι τόσο δύσκολες, ε, τόσα εμπόδια στον δρόμο μπορεί να είναι πολύ απογοητευτικό. Και μην ξεχνάμε ότι, ότι όταν ο κύριος Λάτιμερ το 2000 ε, έκανε αυτή την αναφορά για το τι συνέβαινε στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο βασικός του στόχος, η βασική του ανησυχία ήταν η ποιότητα του νερού που τα παιδιά του, τα εγγόνια του και τα άλλα παιδάκια ε, είχαν στη διάθεσή τους για να κολυμπήσουν. Αυτός βρισκόταν πάνω από τα βράχια στο Whitburn κοιτούσαν δηλαδή ουσιαστικά τα σημεία διαρροής. Είχαν τη μοναδική, μια μοναδική ας πούμε, ένα, ας πούμε πλεονέκτημα ε, να βλέπουν οι δύο σώμαση πώς ε, συνέβαιναν αυτές οι διαρροές. Και θέλω να καλέσω και τα μέλη της Επιτροπής να επισκεφθούν το τόπο αυτό, γιατί πραγματικά βλέπουν με τα μάτια τους τι σημαίνει σε αντιδιαστολή με τα επίσημα στοιχεία. Πραγματικά είναι αυτά τα φαινόμενα αυτά, αυτά που λένε οι ακτιβιστές. Χρειά, χρειάστηκαν πάρα πολλά χρόνια για να φτάσει η υπόθεση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ε, και να εξεταστεί από αυτό. Χάρη στην ε, πολλή δουλειά που έκανε ο Στίφεν Γιούς, ε, ο πρώην Ευρωβουλευτής από, για τα Βόρειο Ανατολικά και Χάρη σε αυτέ τι προσπάθειε έφτασε αυτή η πρότυπη υπόθεση στο δικαστήριο. Ε, δεν θέλω να υποτιμήσω το τι έχει γίνει μέχρι τώρα. Το πρόβλημα είναι ότι τα νερά τη Νοθάμπρια, ε, ή μάλλον έπρεπε η περιοχή της Νοθάμπρια ε, μέσα σε πέντε χρόνια να εφαρμόσει την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Τώρα, τους δόθηκε μια επιπλέον περίοδος ε, χάρης για να συμμορφωθούν και μόνο την τελευταία μέρα της λήξης της περίοδου χάριτος ε, συμμορφώθηκαν, ας πούμε. Ήταν μια πολύ μακρά ιστορία και χάρη σε αυτό. Και επειδή ε, οι κάτοικοι ακόμα παίρνουν φωτογραφίες ε, που αποδεικνύουν ότι στα βράχια, εκεί στις λιμνούλες στα βράχια ε, υπάρχουν ε, ανεπεξέργαστα λύματα και απόβλητα, ας πούμε, υπάρχει πάρα πολύ ε, δυσπιστία. Εγώ αυτό που λυπάμαι ως Ευρωβουλευτής είναι ότι δεν κατάφερα και σε άλλες αναφορές να φέρω όλους τους συμμετέχοντες σε ένα τραπέζι, ούτω ώστε να βρεθεί μια καλή λύση στην κατάσταση αυτή. Αλλά κάνω έκκληση στην Επιτροπή να προσπαθήσουν να οργανώσουν μια τέτοια συζήτηση στρογγυλή τραπέζης, να έρθουν σε επαφή με την τοπική κοινότητα, από την οποία προέρχεται και ο κύριο Λάτιμερ, γιατί θα ήταν τραγικό εάν παλεύαμε για αυτή την περιβαλλοντική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με επίμονους ε, ε επιτόπου που θέλουν να εφαρμοστεί αυτή η νομοθεσία και θέλουν να βελτιώθει το περιβάλλον στις κοινότητές τους και παρόλα αυτά δεν εφαρμόζεται, υπάρχει δυσπιστία και η νομοθεσία αυτή δεν φέρνει τα αποτελέσματα που θα έπρεπε να φέρει στι κοινότητε αυτέ. Το τελευταίο σημείο είναι να επαναλάβω αυτό που είπε ο κ. Λάτιμερ, ότι υπάρχει μία αμφισβήτηση για τα δεδομένα, για, τα, για τι διαρροέ, τον αριθμό των διαρροών και την ποιότητα του νερού και τα, τα δεδομένα για την ποιότητα του νερού στην παραλία. Και ενθαρρύνω την Κομισιόν αναγνωρίζοντας βέβαια το, τα περιθώρια έρευνας που έχει η Κομισιόν, να, να επαληθεύσει ανεξάρτητα από τα δεδομένα, ανεξάρτητα από αυτά που τους λένε οι Βρετανικές αρχές, για να δουν η δίσο μας ποια είναι η κατάσταση στην περιοχή αυτή. Ελπίζω τελικά ότι το Brexit... Κοιτάξτε, εγώ είμαι υπέρ του, της παραμονής, έτσι. Ε, πιστεύω ότι θα έπρεπε να είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι μόνο για περιβαλλοντικούς λόγους, αλλά για πολλούς λόγους ε, και για το καλό της βορειοανατολικής Αγγλίας. Ε, τουλάχιστον ιδανικά σε μια μεταβατική περίοδο ε, να παραμείνουμε μέλος και να ε, εφαρμοστούν όλοι αυτοί οι κανόνες. Εγώ θα ήθελα η περιβαλλοντική νομοθεσία να εφαρμοστεί και, και στο επέκεινα. Δεν θα πρέπει να θεωρηθεί το Brexit η ευκαιρία για να χαλαρώσουμε τις προσπάθειες και να μην εφαρμόσουμε την ευρωπαϊκή νομοθεσία σε περιοχές όπως ε, η εκλογική μου περιφέρεια. Γιατί μιλάμε για περιοχές όπου ο κόσμος έχει γίνει κοινικός, όπου ψήφισε υπέρ του Brexit, ε, όπου ε, υπάρχει πρόβλημα, ας πούμε. Εδώ πραγματικά μπορούμε να δείξουμε την αξία της συμμετοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στους ντόπιου, στις κοινότητες αυτές στο Whitburn και σε περιοχές ε, βόρεια από το Sutherland. Ευχαριστώ, Τζουντ. Πραγματικά βλέπω ότι είναι ανάμεικτα τα συναισθήματα, γιατί δεν ξέρουν οι άνθρωποι τι θα χάσουν ε, να είναι μέρος της προστασίας του περιβάλλοντος, ε, είναι και με τις αρετές της ε, συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριος Γιάρ. Yeah, <clears throat> Bei dieser Petition äh, liegen die Fakten ja offen. würde sagen... Λοιπόν, ε, νομίζω ότι πρέπει να διατηρήσουμε ανοιχτή αυτή την αναφορά και να αφήσουμε τη δυνατότητα στην Επιτροπή να δράσει. Και καθώς ε, έρχεται από το Ηνωμένο Βασίλειο η αναφορά αυτή και κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει τις επόμενες εβδομάδες, ε, καλό την Επιτροπή να δράσει τώρα. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει στις 29 Μαρτίου ή τι δεν θα γίνει αλλά μην σκέφτεστε σαν να έχει ήδη βγει το, Ευρω... το Ηνωμένο Βασίλειο και δεν έχει κανένα νόημα να αναλάβουμε δράση από αυτού. Όχι, εγώ προτείνω να ακολουθήσουμε την ε, τακτική διαδικασία, να διατηρήσουμε ανοιχτή αυτή την αναφορά και να συνεχίσει η Κομισιόν της Εργασίας της ε, και η Επιτροπή και ίσως σε κάποιες εβδομάδες να έχουμε μια μεγάλη έκπληξη και μπορεί και οι Βρετανοί φίλοι μας ε, να μας συντροφεύσουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Πρόεδρος, νομίζω ότι συμφωνείς μαζί μου, Τσουτ. Ο κύριος Τερικάμπρας, καταρχήν. Συμφωνώ απόλυτα Νομίζω ότι είναι ένα ευρωπαϊκό ζήτημα. Φυσικά υπάρχουν κάποια τεχνικά ζητήματα σημαντικά που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν και να επιληθούν. Είναι ενδιαφέρον να ακούμε ότι υπάρχουν αρκετές καταγγελίες, όχι μόνο του κυρίου Λάτιμερ. Και ότι έχουν ε, υπάρξει βελτιώσεις ε, στο σύστημα συλλογής ε, των υδάτων που όμως δεν είναι ικανοποιητικές. Νομίζω ότι θα πρέπει να υποστηρίξουμε την Κομισιόν να ξεκινήσει η διαδικασία επί παραβέση και θα πρέπει να υποστηρίξουμε και τον κύριο Λάτιμερ στα αιτήματά του που είναι δίκαια και κατάλληλα. Είμαι λοιπόν υπέρ του αναφέροντος. Πολύ ωραία. Και τώρα θα συνοψίσω εγώ. Θα διατηρήσουμε ανοιχτή αυτή την αναφορά. Θα περιμένουμε την, να ενημερωθεί η Κομισιόν και να συνεχίσει το διάλογο με τις Βρετανικές Αρχές ε, για το πώς αντιμετωπίζουν αυτό το μεγάλο όγκο απορρίψεων ε, στο Whitburn και νομίζω ότι πρέπει να στείλουμε και μια επιστολή στις αρχές του Ηνωμένου Βασίλειου ω επιτροπή. Δηλαδή ότι συνεχίζουμε να ενδιαφερόμαστε και να τους γνωστοποιήσουμε ότι παρακολουθούμε το ζήτημα για να δούμε τι κάνουν με αυτό το θέμα της επεξεργασίας των λιμάτων. Και επίσης η Κομισιόν, την Κομισιόν την παροτρύνουμε να συνεχίσει την καλή δουλειά και ελπίζουμε να επιληθεί το ζήτημα αυτό άπαξ και το συντομότερο. Και στον κύριο Λάτιμερ ε, παρακαλώ Τζούντε να του διαβιβάσει τις ευχές μας για ταχεία ανάρρωση. Ωραία, ας προχωρήσουμε στο επόμενο θέμα που αποτελεί ε, την, το follow-up της ερευνητική επίσκεψης στη Γαλλική που έλαβε χώρα το 2013 πριν ξεκινήσει καν αυτή η θητεία. Εγώ δεν ήμουν μέλος αυτής της επιτροπής, αλλά παρόλα αυτά έλαβε χώρα αυτή η αποστολή. Υπήρξαν κάποιες συστάσεις και νομίζω ότι αυτό που τώρα μπορούμε να κάνουμε είναι να αντικατοπτρίσουμε ε, σε τι συνίστατο η αποστολή και ποιες ήταν οι συστάσεις της Επιτροπής. Να δώσω το λόγο καταρχήν στους αναφέροντες. Ε, είναι ο κύριος Ρεγέρα Γόμες και ο κύριος Φελίπε Κανός Εντονάδο. Έχετε ο καθένας 4-5 λεπτά, όμως αν είστε σύντομοι τόσο το καλύτερο. Hola, buenas tardes. En principio... Eh, Καλησπέρα σας. Χαίρομαι για αυτή την ευκαιρία που μου δίνετε για να σας υπενθυμίσω το πρόβλημα ε, που έχουμε στη Ρία Δελμπούργκο, σε αυτά τα φιόρδα, ε, στον ποταμόκορπο αυτό, ε, που ξεκίνησε πριν από πέντε χρόνια. Η Ρία Δελμπούργκο στην Ακορούνια ήταν ένα φιόρδ ε, με μεγάλο δυναμικό ε, παραγωγής οστρακοειδών, όπως το αποδεικνύει το γεγονός ότι στη δεκαετία του 90 είχαμε περίπου 2.167 ηχθειοκαλλιεργητές ε, και καταγεγραμμένους ηχθειοκαλλιεργητές, ενώ σήμερα είναι πολύ λιγότεροι λόγω της πολύ μεγάλης μόλυνσης που έχει προκληθεί από εκατοντάδες απορρίψεις ανεξέλεγκτες ε, παραδείγματος χάρη ε, αστικά και βιομηχανικά απόβλητα από εταιρείες όπως το σφαγείο Φρικόσα η ε, εταιρεία ε, Ελέον Μπούχε εταιρεία λιπασμάτων κτλ. Μετά από πολλά χρόνια αγώνα από την πλατφόρμα άμυνας της Ρίας Δεμπούργο και της συντεχνίας των αλλιέων της Ακορούνια, ε, εγώ ως εκπρόσωπος της ε, συντεχνίας ήρθα εδώ πέρα για να σας παρουσιάσω ε, το πρόβλημα λόγω της έλλειψης θέλησης από τις τοπικές αρχές, την αυτόνομη κυβέρνηση, την ισπανική κυβέρνηση κτλ. Το πρόβλημα είναι σοβαρό, κοινωνιοοικονομικό και περιβαλλοντικό. Έχουμε το ευρωπαϊκό πλαίσιο, την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης η οποία θα πρέπει να εφαρμοστεί ε, και να... Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να γίνουν, ε, γίνει επεξεργασία των υδάτων, ε, τα οποία στέλνονται και αυτή η νομοθεσία τέθηκε σε ισχύ το 2015. χάρη στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία η ποιότητα των υδάτων βελτιώθηκε αλλά όμως δεν λύθηκε το πρόβλημα της καλλιέργειας ε, οστρακοειδών. Ε, λόγω του γεγονότος έχουμε ε, πάρα πολλές ανεξάρτητες απορρίψεις ε, υδάτων στο φιόρδο αυτό, με πάνω από 300.000 κυβικά μέτρα ηλίως μολυσμένης που έχουν κατεθεί στο βυθό των θαλάσσιων, στους θαλάσσιους βυθούς, λόγω αυτών των οργανικών και χημικών αποβλήτων. Με αυτή την έγινε μια έκθεση και ζητήσαμε, ζήτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από την κυβέρνηση της Ισπανίας να μην φυστεί ούτε κόστους ούτε χρόνου ε, προκειμένου να καθαρίσει την περιοχή αυτή. Ε, ξεκίνησε μια προσπάθεια, ε, φτιάχτηκε ένα σχέδιο καθαρισμού της Ρίας Δελμπούργο πέρασαν πάνω από πέντε χρόνια από τότε που ζητήσατε εσείς από την Ισπανική κυβέρνηση να καθαρίσει την περιοχή και παρόλα αυτά Μέχρι σήμερα αυτό το project δεν έχει ολοκληρωθεί και δεν προβλέπεται ούτε βραχυπρόθεσμα ούτε μεσοπρόθεσμα να εγκριθεί, ούτω ώστε να δοθεί η άδεια από την ε, Ισπανική κυβέρνηση για να γίνουν τα απαραίτητα έργα, ούτω ώστε το φιόρτο δικό μα ε, στη Γαλλικία να ε, καθαρίσει από την μολυσμένη ύλη που επηρεάζουν την χλωρίδα και την πανίδα, τους ηχθειοκαλλιεργητές και τον πληθυσμό που θέλει να ζήσει σε ένα καθαρό και υγιεινό περιβάλλον. Ε, δυστυχώς το 2012 ένα παιδί ε, πέθανε, ε, μπερδεύτηκε εκεί, πιάστηκε στην ε, ηλία αυτή και δεν μπόρεσε να φύγει πριν να ανέβει η παλήρια και πνίγηκε. Όλα αυτά ε, δείχνουν την έλλειψη πολιτική βούληση τη Ισπανική κυβέρνηση και τη αυτόνομη κυβέρνηση τη Γαλλικία να λύσουν το πρόβλημα. Γι' αυτό ήμασταν υποχρεωμένοι να επανέλθουμε εκ νέου εδώ, ούτω ώστε εσεί ε, να κάνετε ό,τι μπορείτε, ούτω ώστε ε, εμεί, οι πάνω από 600.000 κάτοικοι της ε, Μητροπολιτική Περιοχής τη Κορούνια να μπορέσουμε να δούμε για ποιο λόγο η Ισπανική κυβέρνηση, παρά το γεγονός ότι τη ζητήσατε να βελτιώσει το περιβάλλον, δεν έχει κάνει τίποτα. αυτά και ευχαριστώ. Thank you very much, Κύριε Κανός Εντοναδο. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ την ε, Επιτροπή που μας δίνει τη δυνατότητα να παρέμβουμε ε, στην αίθουσα αυτή ως πλατφόρμα για την υπεράσπιση της Ρίας ε, του Βίγκο και θέλουμε να σας παρουσιάσουμε όπως ε, βλέπετε στις ε, διαφάνειες προκειμένου όλοι όσοι είστε εδώ να δείτε πώς κατανέμεται ο πληθυσμός ε, στη Ρία του Βίγο. Έχουμε πάνω από 400.000 κατοίκους. Το Βίγο είναι η κύρια ε, πόλη, 300.000, Ροντοντέλ 29.000, Κάνγκας 26.400, Τονιγρά 17.700, Μπαγιώνα 12.100, μαγιόρ 7.000 και Βιαμπόα 6.000. Στη δεύτερη διαφάνεια θέλουμε να δείξουμε τα πιο σημαντικά σημεία των απορρίψεων σε ολιτηρία. Και δεν είναι τα μόνα σημεία αυτά. Αυτό θέλουμε να το ξεκαθαρίσουμε, αλλά είναι τα μεγαλύτερα. Τα πιο σημαντικά σημεία. Στην τρίτη διαφάνεια βλέπετε κάποιες φωτογραφίες από διάφορα σημεία απορρίψεων και πάλι δεν έχουμε το σύνολο εδώ των σημείων είναι κάποια από αυτά και αν τα συγκρίνουμε, γιατί εμείς λειτουργούμε ως πλατφόρμα με φωτογραφίες που έχουμε από 10 χρόνια πριν, ακριβώς είναι τα ίδια τα σημεία αυτά, 10 χρόνια μετά. Έτσι, λοιπόν, τα μέτρα που έχουν ληφθεί και προτάθηκαν από την Επιτροπή Αναφορών δεν έχουν υλοποιηθεί με αποτελεσματικότητα. Συνεχίζουν λοιπόν να υπάρχουν προβλήματα σε ό,τι αφορά την ποιότητα του ύδατος στη Ρία Δεβίγο. Και από την ποιότητα αυτή του ύδατος ε, έχουν ε, εξαρτηθεί 15.000 θέσει εργασία, ε, αλληλείς και καλλιεργητές μαλακίων, οι οποίοι οδηγήθηκαν οι οποίοι υπέστησαν συνέπειε λόγω τη αλλαγή τη ποιότητα των υδάτων. Στην τέταρτη διαφάνεια βλέπουμε ότι έχει κατασκευαστεί νέο βιολογικό καθαρισμό στο Βίγο που έχει ικανότητα από ό,τι μας λένε για να καλύψει 800.000 κατοίκους, ενώ η πόλη του Βίγα έχει περίπου 300.000 κατοίκους. Το πρόβλημα είναι ότι όταν σχεδιάστηκε αυτός ο βιολογικός ε, καθαρισμός δεν ε, ελήφθης, ε, δεν ελήφθηκαν υπόψη το εξή. Ε, τι υπήρχε πριν, δηλαδή οι υπόνομοι που οδηγούν το νερό ε, στον βιολογικό καθαρισμό και δεν ελήφθη αυτό υπόψη παρόλο που η πλατφόρμα αυτή είπε με κάθε μέσο σε όλες τις ενεχόμενες δικήσεις ότι θα υπήρχε πρόβλημα γιατί κανένας βιολογικός καθαρισμός δεν θα μπορούσε να καθαρίσει όλα τα ύδατα. Γιατί δεν έχουμε ξεχωριστούς σωλήνες για τα όμβρια ύδατα και ξεχωριστούς ε, για τα λίματα. Ε, και ακόμη και όταν δεν βρέχει, υπάρχουν ε, πάρα πολλά υπόγεια ποτάμια, τα οποία χύνονται πρώτα στη Ρία, ενώ σήμερα έχουν διοχετεύσει αυτά τα ποτάμια σε αυτούς τους σωλήνες. Επομένως, κανένας βιολογικός καθαρισμός δεν θα είναι σε θέση να καθαρίσει όλα αυτά. Και μάλιστα αυτός ο βιολογικός καθαρισμός έχει ικανότητα εισόδου νερού 12 κυβικών μέτρων ε, το δευτερόλεπτο, 2,6 ε, ε, κυβικών μέτρων το δευτερόλεπτο είναι ο μέσος όρος της ροής του νερού. Παρ' αυτά, εδώ βλέπουμε μία ικανότητα εκένωση 8 κυβικών μέτρων το δευτερόλεπτο. Δηλαδή τι θα γίνει σε περίπτωση που ο βελικό καθαρισμό δεν μπορέσει να καθαρίσει 12 κυβικά μέτρα. Τι θα γίνουν ε, αυτά τα υπόλοιπα κυβικά μέτρα. Και τέλος ε, πρέπει να πούμε ότι όταν βρέχει το νερό που μπαίνει στους σωλήνες πολλαπλασιάζεται από 20 έως 60 φορές ε, από την κανονική ροή. Δηλαδή, τα 12 κυβικά μέτρα θα μπορούσαν να μετατραπούν σε 80, 60, ανάλογα με την ποσότητα του νερού ή και παραπάνω. Αυτό το λέμε έτσι ώστε εσείς να συνειδητοποιήσετε όλες αυτές τις πτυχές. Στην επόμενη διαφάνεια Θέλουμε να τονίσουμε τι γίνεται με τα αντιλιοστάσια. Εδώ έχουμε κάποιες αντλίες, ε, στέλνουν το νερό προς το βιολογικό καθαρισμό και κατά μήκος της ακτής του Βίγου υπάρχουν πέντε τέτοια αντιλιοστάσια και αυτά ανοίγουν όταν υπάρχουν ε, πάρα πολύ νερό, ανοίγουν οι πόρτες και υπάρχουν κατευθείαν απορρίψεις στη θάλασσα. Στην επόμενη διαφάνεια, γιατί πιέζει ο χρόνος θα δείτε τον κοινωνικό αντίκτυπο στο περιβάλλον όλων αυτών των απορρίψεων. Δηλαδή εδώ μπορείτε να πάρετε μια ιδέα. Θα μπορούσα άπειρα τέτοια έγγραφα να σας παρουσιάσω. Όλα αυτά θα μας προκαλούσαν μεγάλο πονοκέφαλο. Και στην πρώτη τελευταία διαφάνεια θέλουμε να απευθύνουμε μια έκκληση σε όλους έτσι ώστε η Ρία του Βίγκο, όλε αυτέ τι φωτογραφίε που βλέπετε εδώ είναι βιοπικιλότητα που υπάρχει στη Ρία του Βίγκο. Ένα μέρο τη βιοπικιλότητα και για να τα προστατεύσουμε όλα αυτά και να τα διατηρήσουμε, θα πρέπει να καθαρίσουμε όλα τα νερά όπω πρέπει. Διαφορετικά όλα αυτά θα ξεφανιστούν. Και τέλο, θέλουμε να απευθύνουμε μία έκκληση ως πλατφόρμα και να σας εξηγήσουμε ότι εμείς ως πλατφόρμα συμμετέχουμε στην προστασία της ΡΙΑ και απλώς ζητάμε και περιμένουμε από τους κυρίους βουλευτές και εσείς ε, να εμπλακείτε και να απευθυνθείτε στις αρμόδιες ισπανικές αρχές προκειμένου να ε, θέσουν σε εφαρμογή την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα να ακούσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον κύριο Φερνάντες Γκόμες. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Κομισιόν κατέγραψε όλα αυτά τα ε, σχόλια των αναφερομένων. Θα αναλύσουμε αυτές τις πληροφορίες και όλες τις άλλες πληροφορίες που θα μας στείλετε για να δούμε εάν υπάρχει κάποια παράβαση απέναντι στις υποχρεώσεις που έχει η Ισπανία λόγω της ε, ενωσιακής νομοθεσίας είναι στη διάθεση της Επιτροπής σας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και θα επικοινωνήσουμε. Ευχαριστώ. Οι βουλευτές, η Άννα Μιράντα πρώτα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι σημαντική η μέρα αυτή για, την, για τις ρίας αυτές. Από το 2013 αυτή η Επιτροπή ε, έκανε μία αποστολή στη χώρα μου. Γι' αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχήν όλους όσους στήριξαν αυτή την αναφορά. Και το γεγονός ότι ξανανοίξαμε την αναφορά αυτή τον Νοέμβριο, ούτω ώστε να έρθουν εδώ οι αναφέροντες, είναι πολύ σημαντική αυτή η αναφορά για τους ποταμόκολπους αυτούς. Είχε μεγάλη απήχηση στη χώρα μου θα ήθελα να χαιρετήσω ειδικά ένα άτομο, τον David Λό, που είναι εδώ, που είναι ο γραμματέας, ήταν ο γραμματέας ε, της αποστολής εκείνη, όταν έγινε η αποστολή το 2013. Πρέπει να υπενθυμίσουμε τη δουλειά που έκανε η Επιτροπή αυτή και όλες οι ομάδες. Μιλάμε για χιλιάδες ανθρώπους ε, που τους απασχολεί αυτό το πρόβλημα. Αυτή η έκθεση που την έχω αναχείρας είναι η τελική έκθεση που κάναμε μετά την αποστολή. Όλοι εμείς συμμετείχαμε, ήμασταν διάφορα μέλη. Ο κ. Γκουλά, ο κ. Γουίστρον και άλλοι ε, που συνέταξαν την έκθεση. Ε, υπάρχουν και διάφορες συστάσεις πολύ σημαντικές που αναφέρει η έκθεση αυτή ε, για, τις, για τους ποταμόκολπους. Χρειάζεται χρηματοδότηση και να δοθεί προτεραιότητα σε project, σε έργα που σκοπό έχουν τον καθαρισμό της περιοχής. Είναι σημαντικό για τους Γαλλικιανούς. Εδώ υπάρχουν διάφοροι Γαλλικιανοί, τους ε, χαιρετίζω. Ε, όλοι μαζί αυτά τα χρόνια συνεργαστήκαμε. Πληροφορίες δόθηκαν το 2015, το 2016, 2017, 2018 στην Επιτροπή. Υπάρχει πραγματική ανησυχία ε, για το γεγονός ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί τα έργα θέλουμε να δούμε τι έχει γίνει και τι δεν έχει γίνει. Καταρχάς, ε, μία από τις συστάσεις ε, της έκθεσης αυτής, που δεν έχει ε, υλοποιηθεί, είναι ότι δεν έχει γίνει ένας απολογισμός. Ούτε η γαλλικιανή κυβέρνηση έχει κάνει ό,τι πρέπει για να κάνει πλήρη καθαρισμό. Ειδικά στην Ρία Δερμπούργο, στην Ακορούνια και στο Βίγο. Θα πρέπει να καθαριστεί όλο το σύστημα αυτό της Γαλλικίας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για να διατηρηθεί το περιβάλλον και να υπάρξει οικονομική ανάπτυξη. Ειδικά στον τομέα της ε, αλίας και της ηχθειοκαλλιέργειας στη χώρα μου. Αυτά τα χρόνια που πέρασαν από την επίσκεψή μας, είδαμε ότι η απασχόληση σε ορισμένε από τι περιοχέ αυτέ έχει μειωθεί πάρα πολύ λόγω τη ε, κακή ποιότητα των νερών στι ρίε αυτέ. Ε, μία από τις ε, δράσεις λοιπόν ε, των συστάσεων είναι να ολοκληρωθεί αυτός ο βιολογικός καθαρισμός. Παρόλα αυτά και παρόλα όσα έχουν γίνει, εξακολουθεί να υπάρχει το πρόβλημα. Στη Ριαντελμπούργο υπάρχει πραγματικό πρόβλημα. Έχουμε μια δεύτερη ευκαιρία και χάρη στην αλλαγή της κυβέρνησης, γιατί η προηγούμενη δεν έκανε τίποτα, να καθαρίσουμε την περιοχή από την ε, λάσπη και να βελτιώσουμε την ποιότητα των ε, ποταμόκολπων αυτού. Ε, έχουμε τα διαρθωτικά ταμεία που μπορούν να βοηθήσουν. Ξέρετε ότι υπάρχει μια ανοιχτή υπόθεση εναντίον της ισπανικής κυβέρνησης για το βιολογικό καθαρισμό. Ευχαριστούμε την ομάδα που πρωταγωνίστησε ούτως ώστε να ξανανοίξει αυτή η αναφορά. Όλες οι ομάδες μας στήριξαν εκτός από μία ε, που δεν ήθελε να ανοίξει ξανά η αναφορά. Πάντως είμαστε σε διαφορετική πολιτική συγκυρία τώρα. Είναι πολύ σημαντικό να ακούσουμε του ε, ετούντες γιατί ήρθαν εδώ λόγω της ε, απογοήτευσης που υπάρχει. Πέντε χρόνια πέρασαν από την αποστολή στις, στην περιοχή αυτή τη Ρία, ε, στους παταμόκολπους αυτούς και τίποτα δεν έγινε, δεν έχουν ε, γίνει αυτά που έπρεπε τέλο πάντων. Ε, έχουμε την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με βάση αυτή πιστεύω ότι πρέπει να δοθεί η συνέχεια, να παρακολουθήσουμε την υπόθεση. Να ολοκληρωθεί ο καθαρισμός της Ρίας, Δελμπούργο και να συμμορφωθούμε με τις απαιτήσεις της οδηγίας πλαίσιο για το νερό. Ε, αν υπάρχει χρόνο, θέλω να μου ξαναδοθεί ο, ε, ο λόγος, ούτως ώστε να πω και άλλα πράγματα, αφού μιλήσουν και άλλοι ε, Ισπανοί ε, επισκέπτες. Αν υπάρχει χρόνος. Ο κύριος Μπλάνκο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να καλωσορίσω τους πολίτες της Γαλλικίας και όσους παρευρίσκονται σήμερα εδώ. Αν και εγώ εκείνη τη στιγμή δεν ήμουν βουλευτής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2013, κατόπιν μιας αποστολής υλοποιήθηκε μια έκθεση που περιλάμβανε μια σειρά εκθέσεων και είχα την ευκαιρία να τις διαβάσω πολύ προσεκτικά σε σχέση με το Βίγο αλλά και με το Ρεγανό Σανσερόλ που ε, συμπεριλαμβάνονταν στην ίδια έκθεση και σε σχέση με τον κολπό του Ομπούργο και πέντε με χρόνια μετά. Δεν αλλάζουν βέβαια τα πράγματα από τη μία μέρα στην άλλη για ένα τέτοιο μεγάλο έργο, γιατί ακόμη και αν ε, είχαν γίνει όλες οι εργασίες αποκατάστασης, δεν στην από τη μία μέρα στην άλλη. Μπορούμε όμως να πούμε ότι βλέπουμε κάποια φωτεινά και κάποια σκοτεινά σημεία για το Βίγο αν ε, και δεν έγινε σεβαστή η προθεσμία για την υλοποίηση και τη θέση σε λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού που έπρεπε να τεθεί σε λειτουργία το Δεκέμβριο του 2015, ε, αυτή τέθηκε σε λειτουργία πέρσι τον Απρίλιο και χάρη και στην ευρωπαϊκή χρηματοδότηση από τα ευρωπαϊκά ταμεία υπάρχει τώρα ένα εργοστάσιο που μπορεί να επεξεργαστεί τα λίματα που αντιστοιχούν στους 800.000 κατοίκους και να αποφευχθούν οι άμεσες απορρίψεις στον ποταμόκολπο όταν έχουμε ισχυρές βροχοπτώσεις. Εγώ ξέρω τον εκπρόσωπο της πλατφόρμας. Ε, ανέφερε κάποια τεχνικά στοιχεία ε, ίσως είστε εμπειρογνώμονας, εγώ δεν ε, γνωρίζω και δεν μπορώ να αναφερθώ στα τεχνικά, όμως ε, ξέρω ότι έγινε ένα τόσο μεγάλο έργο με ένα μεγάλο προϋπολογισμό και έγιναν σεβαστά όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά για να αντιμετωπιστεί η πρόκληση που είχαν ενώπιόν του. Ε, δεν ξέρω αν εσεί μπορείτε να μα πείτε κάποια συμπληρωματικά τεχνικά στοιχεία βάσει τη εμπειρία σα ή βάσει των τεχνικών σα γνώσεων. Όμω, αν μπορούσατε, καλό θα ήταν ε, αυτά να φτάσουν και στο Υπουργείο γιατί όπως σας είπα χρειάζεται χρόνος για τη Ρεγανόσα. Αν και δεν σχολιάστηκε, εγώ έχω την υποχρέωση να την αναφέρω, γιατί ε, στην έκθεσή μας γίνεται αναφορά στη Ρεγανόσα. Οι συστάσεις επέμεναν στην αναγκαιότητα να υπάρχει τακτικός διάλογος με την κοινωνία των πολιτών και με τις αρμόδιες αρχές, ε, να υπάρχει διαφάνεια και παρακολούθηση των δραστηριοτήτων. Πέντε χρόνια μετά η Ρεγανόσα δημοσιεύει μία ετήσια έκθεση στην ιστοσελίδα της για διάφορες πτυχές μεταξύ άλλων και την ε, κοινωνική και περιβαλλοντική δέσμευση του εργοστασίου. Υπάρχει μια ετήσια περιβαλλοντική δήλωση σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και έχει συνεδριάσει ενημέρωση ε, με ενώσει και συλλογικότητε τη περιοχή. Επίση, έχει προωθήσει περιβαλλοντικέ ε, πρωτοβουλίε και ένα συνέδριο το 2018 προκειμένου να υπάρχει αποκατάσταση στην περιοχή και συμμετείχαν ε, και οι διτοκαλλιεργητές ε, του Φερόλ. Σε σχέση με τον ποταμό κόλπο του Ομπούργο συνεχίζονται σοβαρές προσπάθειες ε, προκειμένου να αποκατασταθεί η υποβάθμιση του ποταμόκολπου. Συμφωνώ απόλυτα με αυτή τη συλλογιστική και μετά από ένα καιρό παράλυσης και μετά από την παρουσίαση νέου γενικού προϋπολογισμού αν δεν υπάρχει προπολογισμό ε, και δεν έχουν εγκριθεί οι προπολογισμοί. Κοιτάξτε, πρώτα δεν είχε μαγειρευτεί τίποτα. Όμως, αν δεν εγκριθούν οι προπολογισμοί, εγώ σε σεβάστηκα, συνάδελφε, κυρία Μιράντα, και εσύ, ε, δυστυχώς τείνεις να διακόπτεις τους υπόλοιπου. Και εγώ ε, εργάζομαι. Γιατί μπορούμε να δούμε ε, εδώ ότι όλοι εργαζόμαστε στο Κοινοβούλιο. Κοιτάξτε, εγώ είμαι η πρόεδρος εδώ στην αίθουσα και σας παρακαλώ να σεβαστείτε το χρόνο αγόρευσης. Σας δώσαμε το λόγο και έχετε μακρηγορήσει. Τώρα, ο κύριος Λόπας έχει το λόγο. Σας παρακαλώ, αναφερθείτε στο θέμα της αναφοράς, αλλά μην ξοδεύετε την ενέργειά σας σε συναδέλφους, ε, γιατί δεν θέλουμε τώρα εδώ ισπανική φαρσοκομωδία. Συνεχίστε. Ναι. Κοιτάξτε, εγώ είπα κάτι στη συνάδελφο γιατί με διέκοπτε. Αντί να με κατηγορεί, θα πρέπει να ακούσει. Μετά από χρόνια παράλυσης, άλλαξε η κυβέρνηση της Ισπανίας και παρουσιάστηκε ο νέος προϋπολογισμός, το νέο σχέδιο προπολογισμού την ε, προηγούμενη εβδομάδα ο υπουργό ε, Περιβάλλοντος στη Γαλλικία με τις αρμόδιες αρχές ε, έκανε κάποιες κινήσεις και πιστεύω ότι μπορεί να δοθεί λύση στο πρόβλημα του ποταμόκολπου. Ε, το πρόβλημα είναι ότι η αποστολή που έγινε, οι αποστολέ που έγιναν μέχρι τώρα ε, δεν έλυσαν το πρόβλημα στην, στον ποταμόκολπο. Ε, μιλάμε για έναν προϋπολογισμό 8 εκατομμύρια ευρώ. Στην συνεδρίαση της περασμένη εβδομάδας ε, συζητήσαν για τη δυνατότητα να δοθούν 24 εκατομμύρια ευρώ από κοινοτικά ταμεία, ε, ταμεία για να χρηματοδοτήσουν τις δραστηριότητες βυθοκόρησης πέρα από τα 8 εκατομμύρια τα οποία υπάρχουν ήδη εγγραφή στον προϋπολογισμό. Εάν συμβούν όλα αυτά, ε, η κυβέρνηση, και η κυβέρνηση μάλιστα ανακοίνωσε την πρόθεσή τη να προχωρήσει με αυτές τις δράσεις, ούτως ώστε να λύσει ε, το πρόβλημα μέχρι το 2020. Αυτή είναι η δέσμευσή τη. Υπάρχει μια δυνατότητα για να δοθεί οριστική λύση ε, στον ποταμόκολπο. Fine. Now I need to, to actually have put a deadline because we are Τώρα πρέπει να βάλουμε προθεσμία. Δύο λεπτά στη Ροζα και μετά στην κυρία Εύη. Αφού... Mr. Milan, Milan before. Ο κύριος Μιλάν, παρακαλώ. Ελπίζω να είστε ευέλικτοι, γιατί δώσετε τόσο χρόνο στους προηγούμενους ομιλητές. Γιατί να με κόψετε μένα στα δύο λεπτά. Ζητώ η συμμεταχείριση και ευελιξία. Λοιπόν, εγώ εγώ ήμουν ε, μέρο ε, τη αντιπροσωπεία τη Επιτροπή Αναφορά το 2013 και έχω προσωπική και πολιτική δέσμευση για τον καθαρισμό των ποταμόκολπων. Αλλά νομίζω ότι και η δημόσια Δίκηση τη Ισπανία αλλά και τη Γαλλικία ε, και οι Δήμοι έχουν αναλάβει αυτή τη δέσμευση και θεωρώ ότι το αποτέλεσμα, αν δούμε το ισοσύγιο τα τελευταία 20 χρόνια είναι θετικό. Δηλαδή τι γίνεται στις παραγωγικές περιοχές ε, των μαλακίων ε, και έχουμε δει βελτίωση τα τελευταία 10 ε, χρόνια. Σήμερα νομίζω έχουμε φτάσει στο 20% Οι περιοχές που ήταν στο 80 κάτι, μάλλον 60 κάτι, τώρα έχουν φτάσει στο 80 κάτι και οι ζώνες γάμα που ήταν οι χειρότερες πρέπει να έχουν φτάσει ήδη στο 6-7%. Έτσι λοιπόν είναι πολύ μεγάλες οι βελτιώσεις. Εγώ δεν θα έλεγα ότι είναι αρνητικό το ισοζύγιο όσα να έγιναν τα τελευταία χρόνια. Μάλιστα, θετικό είναι το συζύγιο. Βέβαια, δεν μπορεί να αρνηθεί κανεί τα θετικά αποτελέσματα, αν και μένουν πολλά να γίνουν. Τώρα, για την ποταμόκολπο του Βούργο. Είναι σίγουρο ότι πρέπει να γίνει η βυθοκόρηση της λάσπης, όμως δεν υπήρχε παράλυση. Χρειάστηκαν μελέτες, γιατί μια τέτοια βυθοκόρηση δεν μπορεί να γίνει μέσα σε 15 μέρες. Πρέπει να γίνουν μελέτες αντικτύπου κτλ. Και όπως είπε ο κ. Μπλάνκο πριν λίγο, ακόμη, νομίζω την περασμένη ε, τρίτη είχαμε σημαντική ε, συνεδρίαση όπου συμφώνησε επιτέλους η κεντρική κυβέρνηση σε ένα ποσό 8 εκατομμυρίων ευρώ για να γίνει αυτή η βυθοκόρηση. Όμως ε, και πριν είχαν γίνει πολλά στον ποταμό Κολπότομπουργκ. Είχαμε τη διεύρυνση του βιλικού καθαρισμού, είχαμε ένα σχέδιο γενικής αποκατάστασης του ποταμό Κολπού και όταν είχαμε ξηρή περίοδο λειτουργούσαν οι υπόνομοι αλλά και σε περιόδου βροχή Βέβαια δεν σταμάτησε η δίκηση και υπήρχαν, σημείωθηκε πρόοδο. Τώρα για το Βίγο νομίζω ότι δεν μπορούμε να αρνηθούμε το πόσο σημαντικό είναι ο βιολογικό καθορισμό του Λαγάρες. Είναι ένα από ε, τα πιο σημαντικά υδραυλικά έργα ε, της Ευρώπης. Ε, είχαμε πάνω από 200 εκατομμύρια ευρώ που επενδύθηκαν. Φυσικά είχαμε και ευρωπαϊκά κονδύλια και νομίζω ότι άρχισε να λειτουργεί το 2017. Πρόκειται για ένα τεράστιο φαρανικό έργο με πολύ μεγάλη σημασία και φυσικά είναι θετικό το για θετικός υπολογισμός των τελευταίων ετών. Βέβαια, στην του Μπούργκο δεν αρκεί η πρόοδο, γιατί πρέπει να υπάρχει εξυγίανση με την αφαίρεση της ηλίω. Όμως δεν συμφωνώ με αυτήν την τόσο αρνητική εικόνα. Εγώ έχω θετική εικόνα. Θεωρώ ότι υπάρχουν κρεμή πράγματα, όμως η εξυγένση των υδάτων δεν είναι κάτι που γίνεται σε λίγα χρόνια και αυθορμήτω. Χρειάζεται πάρα πολύ καιρό ε, για να γίνουν αυτά τα έργα, αλλά δεν υπήρχε παράλυση από καμία δίκηση, ούτε σε επίπεδο αυτονομία, ούτε σε επίπεδο κεντρική δίκηση. Ε, και αναφέρομαι στα βήματα που έγιναν τα τελευταία χρόνια με κτίρια του Ομπούργο. Και επίσης ακόμα δεν έχουμε προβεί στη φιδοκόρηση της ήλιος, όμως υπάρχει πρόοδος, τη βλέπουμε και γενικά αυτό μπορούμε να το δούμε σε όλα τα ύδατα της Γαλλικίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Δεν μας μένει πια πολύς χρόνος. Σας το λέω ειλικρινά. Τώρα το λόγο ας λάβει η Ρώσα. Όμως, παρακαλώ, όλοι οι Ισπανοί συνάδελφοι, μην παραλάβετε τα όσα ήδη έχουν αναπτύξει οι άλλοι συνάδελφοί σας. Ρώσα, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε όλες ε, οι διοικήσεις, όλες οι αρχές και κυρίως η αυτόνομη κυβέρνηση ε, πήρα, ανέλαβαν δέσμευση για να βελτιώσουν την ποιότητα των νερών. Και οι προσπάθειες αυτές, ε, χάρη σε επενδύσεις που έχουν γίνει, βοηθούν στην εξυγίαση. Από το 2009... 60% και των νερό, δεν ήταν, το νερό δεν ήταν καθαρό, ενώ τώρα έχουμε πολύ περισσότερα καθαρά νερά. Υπάρχει μια βελτίωση από το 2009 ε, πάνω από 10% ε, σε ό,τι αφορά την ποιότητα των νερών. Ε, σε ό,τι αφορά την, τον ποταμόκολπο του Μπούργου, όπως είπε και ο συνάδελφος, επενδύθηκαν πάνω από 200 εκατομμύρια ευρώ και συμμετείχαν εδώ πέρα και οι διάφορες τοπικές αρχές, η αυτονομία, η αυτονομική κυβέρνηση και ευρωπαϊκά κονδύλια. Υπάρχουν χιλιάδες κάτοικοι 600.000 κάτοικοι ε, και χάρη σε όλα αυτά, στις ε, προσπάθειες των αρχών, ε, γίνεται προσπάθεια για να σεβαστούμε την κοινοτική νομοθεσία. Τώρα, για τον ποταμό του ε, έχουν γίνει πολλά πράγματα. Δεν υπήρξε παράλυση, το είπε και ο Πάκο. Ε, έγιναν ε, βελτίωση, έγινε βελτίωση των, ε, του αποχαιρετευτικού συστήματος. Έχουν επενδυθεί πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ για την, ε, τον βιολογικό καθαρισμό, για την εξυγίανση. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για αδράνεια. Είναι θετική η κατάσταση. Υπήρχε μια δέσμευση από τις αρχές και στις 15 του μηνός θα γίνει η συνεδρίαση του Υπουργείου Οικολογικής Μετάβασης και των αυτόνομων φορέων για να γίνει ε, επένδυση 46 εκατομμύριων ευρώ ε, για να επιληθεί το πρόβλημα. Η αποστολή έδωσε καρπούς, ε, οι κυβερνήσει ασχολούνται, δεν είναι πολιτικό το θέμα, ας μην του δώσουμε πολιτική διάσταση, είναι λάθο αυτό. Το περιβάλλον για όλους. Δεν ούτε του Πάκο, ούτε τη της Μιράντα, ούτε κανενός ε, αν σκεφτόμαστε τι εκλογέ το Μάιο και δεν νομίζω ότι θα βοηθήσουμε του κατοίκου και τον ποταμόκολπο. Το βασικό είναι να ε, υλοποιήσουμε τι δεσμεύσει την ε, δέσμευση και τη αυτόνομη κυβέρνηση και τη ισπανική κυβέρνηση. Ε, το βασικό είναι λιγότερη πολιτική, περισσότερη δουλειά. Σα ευχαριστώ πολύ και ιδίω που τηρήσατε το χρόνο σα. Η Εύη. Είμαι πολύ σύντομη. Ήθελα το λόγο. Ήθελα να παρέμβω για αυτές τις αναφορές για να υποστηρίξω τα αιτήματα των αναφερόντων αλλά και τη συνάδελφο Μιράντα. Και να υποστηρίξω και την έκθεση της Επιτροπής πριν πεντέτη, γιατί θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικός ο ρόλος των αναφερόντων και των υπογεγραφόντων να συνεχίζουν να προωθούν τη δημόσια συζήτηση και την επαλήθευση της σωστής εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας, γιατί οι πολίτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν και γι' αυτό το λόγο το δικαίωμα της υποβολής αναφοράς για να πιέσουν έτσι ώστε το κράτος μέλος να μπορεί να σεβαστεί την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία πλήρω. Εγώ νομίζω ότι τα βήματα που έγιναν ε, ήταν ε, πολύ αργά γιατί πέρασαν πάρα πολλά χρόνια και το πρόβλημα συνεχίζει να υπάρχει. Πρέπει να δοθεί μια περαιτέρω όθεση γιατί το αξίζουν οι πολίτες, το αξίζει και το περιβάλλον όπου ζούμε, που δυστυχώς το κακοχειριζόμαστε. Το θέμα των υδάτων ε, είναι ένα σημαντικό θέμα όχι μόνο στην Ισπανία αλλά και στην Ιταλία και θα πρέπει να υπερασπίσουμε αυτό το πόρο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Μητροφάνος. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε που με επιτρέπετε να εκφράσω την άποψή μου. Προ πενταετίας η κυρία Σντάνοκα, προκάτοχός μου, είχε συμμετάσχει στην fact-finding mission στην περιοχή του Βίγο και όταν επέστρεψε συζητήσαμε μαζί της τα αποτελέσματα, τα συμπεράσματα δηλαδή αυτής της αποστολής. Θυμούμε τρία πράγματα που είχε πει. Πρώτο, εγώ ίδιος ανακάλυψα ότι η τοπική κοινωνία είναι έντονα δραστηριοποιημένη για να επιληφθεί των συμφερόντων της, υποβάλλοντας αναφορές στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και καλό παράδειγμα για όλες τις ευρωπαϊκές τοπικές κοινότητες. Δεύτερο, είναι θετικό που η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τόσο υψηλά πρότυπα περιβαλλοντικής προστασίας. Πρότυπα τα οποία εάν εφαρμοστούν μπορούν να αλλάξουν τη ζωή των Ευρωπαίων πολιτών. Και τρίτο, θα δείτε και θα δούμε τα επόμενα χρόνια την επιρροή που θα ασκήσουν αυτές οι έρευνες και το γεγονός ότι επισκεφθήκαμε την ελόγω και ότι η Κομισιόν διαρεύνησε την υπόθεση αυτή. Έχουμε δώσει και κίνητρα και στην κεντρική ισπανική κυβέρνηση αλλά και στις τοπικές αρχές για να επιλύσουν τα περιβαλλοντικά αυτά προβλήματα της περιοχής. Αυτά που βλέπουμε ωστόσο τώρα είναι ότι μετά από μια πενταετία τα προβλήματα δεν έχουν επιληθεί. Εξακολουθούμε να συζητούμε τα ίδια θέματα ποιότητας νερού και ούτω καθεξής. Εγώ υποστηρίζω τους αναφερομένους την ε, τοπική κοινωνία, δηλαδή τις οργανώσεις της τοπικής κοινωνίας και οφείλουμε να, ρωτήσουμε, να ζητήσουμε μάλλον από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει μέτρα, δηλαδή να κάνει βήματα ώστε να προβλεφθούν λύσεις που θα επιτρέψουν να προστατευτούν τα συμφέροντα και δικαιώματα της τοπικής κοινωνίας. Ευχαριστώ. Εσείς κύριε Τερικάβρας. Θα είμαι σύντομος. Δεν θα επαναλάβω τίποτα από αυτά που είπαν οι άλλοι. Ένα λεπτό θέλω. Στηρίζω απόλυτα τον αγώνα σας για τους ποταμόκολπους της Γαλλικίας. Είναι τεράστιο θέμα. Είναι κρίμα, υπήρξαν καθυστερήσεις, πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Είμαστε σε καλύτερο δρόμο τώρα. Μία αμφιβολία έχω, κάτι που με εξέπληξε. Τι με εξέπληξε, η Κομισιόν δείχνει το ενδιαφέρον της μεν, αλλά μοιάζει να μην ξέρει τίποτα. Α, λέει, δεν ξέρουμε τίποτα εμείς. Περιμένουμε πληροφορίες. Έρχεται η Κομισιόν, πάντα όμω για διάφορα θέματα με πολλέ πληροφορίε. Εδώ δεν είχε καμία πληροφορία για αυτό το θέμα. Αυτό με εξέπληξε. Ίσως να μην κατάλαβα κιόλα καλά. Αλλά νομίζω ότι αυτό είπε η Κομισιόν. Δεν είχε πληροφορίε, δεν είχε στοιχεία. Interesting conclusion καταλήγω στο ίδιο συμπέρασμα. Εδώ ολοκληρώσαμε τώρα με την λίστα των ε, μελών που επιθυμούσαν να λάβουν το λόγο. Θα παρακαλέσω πάλι για ένα λεπτό όμως πραγματικά τους αναφερομένους. Ορίστε κύριε. Eh, λοιπόν, να διευκρινίσω κάποια πράγματα. Τα... Ε, δώσαμε κάποια δεδομένα. Οι δικοί μας τεχνικοί, οι οποίοι κάνανε το... που συμμετείχαν στο έργο του βιολογικού καθαρισμού, Μα έδωσαν δεδομένα. Μετά από ένα έτος λειτουργίας του βιολογικού καθαρισμού για το Βίγο, επειδή τους ρωτήσαμε, αναγνώρισαν ότι δεν έχει γίνει τίποτα για το πώς φτάνουν, για τη διαδρομή που κάνουν τα ύδατα μέχρι να φτάσουν στο βιολογικό καθαρισμό. Αυτό δεν ελήφθηκε υπόψη, τη διαδρομή των υδάτων δηλαδή, ε, μέχρι να φτάσουν στο βιολογικό καθαρισμό, κανένα δεν την άλαβε υπόψη. Εάν είχαν γίνει σωστά τα πράγματα, θα, ήταν, ε, θα είχαμε βοηθήσει τον Βίγκο. Ευχαριστώ την Επιτροπή σας, ευχαριστώ τους ε, συντρόφους και θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε διάφορα πράγματα. Εμείς ξέρουμε πολύ καλά ότι για να λύσουμε ένα πρόβλημα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχει. Εάν δεν το αναγνωρίσουμε, δεν θα επιληθεί ποτέ. Αυτό, που, αυτό ακριβώς κάνει οι, όλες οι αρχές στην Ισπανία. Οι αυτόνομες ε, αρχές, οι τοπικές αρχές και οι εθνικές αρχές. Ευχαριστούμε τουλάχιστον ε, εδώ την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που κάνουν κάποια πράγματα. Ξέρω ότι δεν μπορεί να υποχρεώσει τους Ισπανούς. Αλλά αν μας άκουγαν στην Ισπανία, όπως μας ακούτε εσείς, δεν θα χρειαζόταν να έρθουμε εδώ. Δεν θα ερχόμασταν καν εδώ. Δεν μας ακούνε όμως. Η πρόεδρο, σας ευχαριστώ πολύ. Θα θέλατε και εσείς να λάβετε το λόγο. Σας παρακαλώ όμως σύντομα. Θα ήθελα να συμφωνήσω με όσα σχολίασε εδώ ο συνάδελφος, να τονίσω ότι αισθανόμαστε σαν να είμαστε απροστάτευτοι κατά κάποιο τρόπο και ερχόμαστε εδώ να ζητήσουμε τη δική σας προστασία και τη δική σας υποστήριξη. Επίσης να πω ότι θεωρώ υπερβολικό, όσο μεγάλο και αν είναι το έργο, μιλάμε για τα περασμένα πέντε έτη. Νομίζω ότι φτάνει και περσεύει ο χρόνος για να γίνει βυθοκόρηση του ποταμόκολπου του Μπούργκο που παρουσιάζω εγώ τώρα εδώ. Και αν θέλει ο Θεός, θα φανεί και στο μέλλον. Και αν ξεκινήσει το έργο, θα χρειαστεί πολύ λιγότερος χρόνος από όλες αυτές τις προετοιμασίες και τις καθυστερήσεις που βιώνουμε σήμερα. Χωρίς ε, να μακρηγορήσω, θα ήθελα και πάλι να σας ευχαριστήσω που μας δίνετε την ευκαιρία να έρθουμε εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα, θα κάνω μια προσπάθεια να συνοψίσω κάτι που δεν είναι ούτε ιδιαίτερα εύκολο ούτε ιδιαίτερα απλό. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει δώσει ουσιώδη απάντηση. Είδαμε ότι ενώ των βελτιώσεων θα ήταν σωστό να είχαμε λάβει μια ουσιαστική απάντηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αν δηλαδή η επιβεβαίωση ήταν ε, διαφανής και σαφής. Πιστεύω ότι εμείς ως Επιτροπή Αναφορών δεν μπορούμε να κλείσουμε ακόμα τις αναφορές. Πρέπει να τις κρατήσουμε ανοιχτές. και να περιμένουμε έως ότου μας δοθεί αξιόπιστη ενημέρωση για την εξέλιξη όλων των αναφορών. Ενημέρωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και από τις Ισπανικές Αρχές. Άρα αυτό που χρειάζεται να κάνουμε είναι να αποστείλουμε επιστολή και πάλι στις Ισπανικές Αρχές και να υπενθυμίσουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα πρέπει να παραμείνει σε στενή επαφή με τις Ισπανικές Αρχές μέχρι ότου δώσουν επιταγή εν λευκό, ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε καλή την πίστη. Αλλά θα πρέπει να έχουμε αξιόπιστες πληροφορίες μέχρι ότου, ε, μάλλον πριν να κλείσουμε την ε, ε, αναφορά. Μια ερώτηση ε, σε σχέση με τον πενταμόκολπο του Βίγο. Λέει η Κομισιόν, δεν ε, παρακολουθούμε περαιτέρω αυτό το θέμα, γιατί γίνονται σεβαστέ υποχρεώσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση ε, σε όσα λέει η οδηγία για την επεξεργασία των λιμάτων. Η Κομισιόν όμω δεν το έχει πει αυτό. Γιατί αν ε, ισχύει αυτό το έγγραφο, τότε μήπω θα μπορούσαμε να δούμε διαφορετικά τα πράγματα για τον ποταμό του Βίγο. Μου το στείλατε εσεί από την Κομισιόν αυτό το έγγραφο, γιατί εγώ το ζήτησα. Η Πρόεδρος είπε ότι δεν έχουμε πληροφορίε. Εγώ έχω όμως ε, την ε, κοινοποίηση της ε, Κομισιόν. I would like... Η Πρόεδρος. Θα ήθελα τώρα να προσκαλέσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τώρα κοιτάξτε, στην γραπτή σας απάντηση αναφέρεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καταλήξει ότι δεν πρόκειται να παρακολουθήσει περαιτέρω την ε, αναφορά αυτή. Όμως, τα πράγματα στα οποία στηρίζετε τη θέση σας αυτή ανατράπησαν από τους αναφερομένους. Άρα θα πρέπει να τοποθετηθείτε ξανά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πράγματι, η Κομισιόν ε, έχει δημοσιεύσει διάφορες ανακοινώσεις ε, σε σχέση με τις διάφορες αναφορές που συζητήθηκαν εδώ και ξεκάθαρα εκφράστηκε ποια είναι η θέση της Κομισιόν συγκεκριμένα σε σχέση με το φιλικό καθαρισμό του Βίγο η Κομισιόν έλαβε πληροφορίες από τις Ισπανικές Αρχές όπου βεβαιώνεται ότι αυτός ο βιολογικός καθαρισμός λειτουργεί εδώ και πολλού μήνε και έχουν δοθεί και δείγματα ε, από τα ύδατα και επιβεβαιώνεται ότι η επεξεργασία των αστικών λιμάτων συνάδει με την οδηγία επεξεργασία των αστικών λιμάτων. Παρ' όλα αυτά, όλες οι πληροφορίες που παρουσιάστηκαν από τους ε, ε, αναφέροντες δεν ήταν γνωστές στην Κομισιόν, γι' αυτό δεν μπορούμε να τοποθετηθούμε αυτή τη στιγμή μέχρι να μας σταλούν επισήμως. Θα τις αναλύσουμε, θα τις επαληθεύσουμε και θα δούμε αν μπορούν να υπάρχουν νέα στοιχεία που να δείχνουν νέα παράβαση. Όμως, σε σχέση με τον βιλικό καθορισμό του Βίγο, οι πληροφορίες που έχει η Κομισιόν είναι ότι ε, έχουν γίνει σεβαστές οι υποχρεώσεις σε σχέση με το σεβασμό της Ευρωπαϊκή Νομοθεσίας και στις ε, τελευταίες ανακοινώσει για το Μοδομόκολπο του αναφέρεται με σαφήνεια ποια είναι η θέση τη Κομισιόν. Σα ευχαριστώ. I am not intending to give... Δεν προτίθεμαι να ανοίξω και πάλι τη συζήτηση. Θα πράξω το εξή. Ακούσαμε την δήλωσή σα προηγουμένω, την έχουμε και γραπτώσει αλλά οι αναφερόμενοι καταθέτουν νέα στοιχεία. Αυτό σημαίνει ότι εσείς και οι Ισπανικές Αρχές θα πρέπει να διερευνήσετε αν όντως ευσταθούν τα νέα αυτά δεδομένα και να επανέλθετε ώστε να αντιμετωπίσουμε διαφορετικά την αναφορά. Γιατί τώρα τις αναφορές μάλλον. Διατηρούμε ανοιχτέ τι αναφορέ και αναμένουμε ταχεία απάντηση εκ μέρου σα, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να πράξουμε. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστούμε του αναφερομένου οι οποίοι ταξίδεψαν από μακριά από την όμορφη Ισπανία για να έλθουν έως εδώ και σας εύχομαι καλή επάνωδο στις αιστείες σας. Τώρα, ας προχωρήσουμε ε, Δεν μας χειροκροτούν τόσο συχνά εδώ στην Επιτροπή Αναφορών. Σας ευχαριστώ. Τώρα η επόμενη αναφορά είναι η 480 για την προσπάθεια επιτροπής της Πιάτσα Ντάρμι να αποτρέψουν κατασκευή σε ε, οικοδομές, οικοδομική δραστηριότητα δηλαδή, σε ε, πάρκο ή ε, άλλο δημόσιο χώρο. Ο κύριος Προφίλη θα λάβει το λόγο. Θα παρακαλέσω τους Ισπανούς φίλους μας να αποχωρήσουν από την αίθουσα χωρίς συζητήσεις. Αν θέλετε να μείνετε, μείνετε. Ευχαριστώ, αλλά παρακαλώ ήσυχα. Πολύ ευχαρίστως να παραμείνετε. And now, Mr. Profili, the floor. Κύριε Προφίλη, έχετε το λόγο. Καλησπέρα. Λέγομαι Διέγκο Προφίλη και είμαι ο πρώτος υπογράφων της αναφοράς ε, για την υπεράσπιση τη πρώην Πιάτσα Ντάρμι στο Μιλάνο. Μαζί με άλλου εκπροσώπου που είναι παρόντο εδώ, είμαι τμήμα τη Επιτροπή των Πολιτών για την Πιάτσα Ντάρμι, που μαζί με άλλου Μιλανέου πολίτε και την οργάνωση Πάρκο Πιάτσα Ντάρμι, το Πάρκο Πιάτσα Ντάρμι Κυπουρή, προτείνει αυτή την αναφορά για την περιβαλλοντική και ιστορική προστασία αυτού του χώρου. Είναι ένας δημόσιος χώρος που είναι εγκαταλειμμένος τώρα, αλλά που χρησιμοποιούνταν μέχρι 20 χρόνια πριν από τον Ιταλικό στρατό για στρατιωτικές ασκήσεις και γυμνάσια. Έχει μία έκταση περίπου 42 εκτάρια και βρίσκεται στα δυτικά της πόλης, μόνο 5 χιλιόμετρα από το κέντρο του Μιλάνου. Αποτελείται από 35 περίπου εκτάρια πράσινης ε, δασόδους περιοχής και έχει απομονωμένες κάποιες, ε, κάποια στρατιωτικά κτίρια ε, της δεκαετίας του 30 και του 40 του 20ου αιώνα. Ε, στρατιωτική χώρη ήταν αυτή. Ο ιδιοκτήτης που, το Ιταλικό που είναι το Ιταλικό Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών μέσω μιας εταιρεία του, την Invit, ε, που είναι ΑΕ, σκοπεύει να πουλήσει το χώρο σε ιδιώτες. Με βάση το χωροταξικό σχέδιο του Μιλάνου ε, υπάρχει δυνατότητα να οικοδομηθούν περίπου 4.000 ε, κατοικίες, κτίρια, εν πάση περιπτώσει, διαφορετικών σκοπών. Η επιλογή ε, αυτή ελήφθη το 2014 χωρίς καμία δημόσια διαβούλευση με τους Μιλανέζους πολίτες, ούτε, καμία, ούτε μέσω καμία συμμετοχικής απόφασης με τη συμμετοχή των πολιτών. Αυτή η πράσινη περιοχή ε, και το ενδιάτημα αυτό βιοποικιλότητας είναι ε, καρπός μιας ε, αυτόματης, αυθόρμητης διαδικασίας επιστροφής του χώρου στο περιβάλλον που είχε που κράτησε επί Μιλάμε για αστική πράσινη περιοχή με άγρια χλωρίδα και πανίδα, με δάση, με υδροβιότοπους, ε, με έλι και ε, υδρόβια φυτά, ε, βάτραχους και πτηνά, 39 από τα οποία, 39 διαφορετικά πτηνά, 34 από αυτά προστατεύονται από την οδηγία 209-147 και κάποια αμφίβια τα οποία προστατεύονται από την οδηγία ε, για τα ενδιαιτήματα 92-43. Ξέρουμε ότι το Μιλάνο είναι μια πολύ έντονα αστική περιοχή όπου 31,9 τετραγωνικά μέτρα πράσινου αντιστοιχούν σε κάτοικο, ενώ στη Βαρκελόνη 94,6, 133,6 στο Μόναχο, 104 στην Στουτγάρδη κτλ. Ξέρουμε ότι αυτός ο χώρος έχει μεγάλη αξία λόγω της βιοπικιλότητας, αλλά παίζει και ένα σημαντικό ρόλο για να μειωθούν ε, οι ακραίες θερμοκρασίες, τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Έχει σημαντικό, σημαντική επίπτωση στην ποιότητα του νερού, στο υδρογεολογική ισορροπία κτλ. και στην μείωση της ρήμασης, ατμοσφαιρικής Έπαιξε σημαντικό ιστορικό και ανθρωπολογικό και κοινωνικό ρόλο επίσης. Ήταν το πρώτο αεροδρόμιο του Μιλάνου το 2014 και ο μηχανικός Φορλανίνη ε, έφτιαξε το περίφημο πιδαλιούχο αερόστατο. Είχαμε ε, του τους στρατώνες τα Μπάρμπαρα και το ε, νοσοκομείο, στρατιωτικό νοσοκομείο του Μπάτζο. Ε, υπάρχει μια ιστορική μνήμη στους ε, Μιλανέους πολίτες. Πολλές ε, επιτροπές, πολλές ενώσεις, Ιταλοί και ξένοι κινητοποιήθηκαν. Όπως παραδείγματος χάρη το Δημαρχείο 7 η πόλη του Μιλάνου, η Λεγκαμπιέντε, το, ε, η Ένωση Ασώσουμε το Περιβάλλον, η ΛΥΠΟΥ, ε, το WWF. Και αν λάβουμε υπόψη μας την, ε, σύμβαση για, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για, τον, για την Ήπεθρο και τις ευρωπαϊκές οδηγίες για την περιβαλλοντική ευθύνη και διαφύλαξη τόπων διοπικιλότητα, ζητάμε από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να υποστηρίξουν τους φορείς που σας ανέφερα και να ζητήσουν από το Υπουργείο Οικονομικών και Οικονομίας, που είναι ο ιδιοκτήτης και από την, το Δήμο του Μιλάνου, που διαχειρίζεται το χωροταξικό σχέδιο, Ζητάμε λοιπόν η πιάτσα Ντάρμι να διατηρηθεί και να αξιοποιηθεί και να γίνει δημοτικό πάρκο, ε, ένα, ένα φυσικό κεφάλαιο ποικιλότητας και να ταξινομηθεί ως χώρος ειδική προστασίας και για τα πτηνά και για τα αμφίβια. Ζητάμε επίσης το Υπουργείο Οικονομικών και Οικονομίας να επιστρέψει τον τόπο αυτό στο κοινό, σε δημόσια, συλλογική και κοινωνική χρήση και να μην γίνουν όλες αυτές οι επιχειρήσεις από ιδιώτες. Σας ευχαριστώ που μας προσκαλέσατε, ε, που μας δίνετε τη δυνατότητα να συζητήσουμε αυτό το σημαντικό θέμα. Ελπίζουμε ότι η πιάτσα Ντάρμι και χάρη στη συνεισφορά σας θα διασωθεί, ότι θα γίνει ένας νέος ε, δημόσιος ε, τόπος του Μιλάνου, μνημείο φύσης και ιστορίας. Πρέπει να σώσουμε την πιάτσα Ντάρμι. Ευχαριστώ. Thank you very much. Η Πρόεδρο, σας ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ που επενδύσατε χρόνο και ε, τόση ενθουσιώδη δραστηριότητα στο θέμα αυτό. Θα παρακαλέσω τώρα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να φωτίσει περισσότερο το θέμα. Η κυρία Πλούνα, Μανταλένα Πλούνα. Καλό σας απόγευμα κυρία Πρόεδρε και σας ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Πρώτα θα ήθελα να ευχαριστήσω τους αναφερομένους για τις ε, παρεχόμενες πληροφορίες και για τα έγγραφα που συνδέουν την αναφορά, που συνοδεύουν μάλλον την αναφορά. Θα αξιολογήσουμε τις πληροφορίες που περιέχουν τα έγγραφα και θα υποβάλουμε ε, γραπτή κοινοποίησή μας το δυνατόν συντομότερο στην Επιτροπή Αναφορών. Για την ώρα θα ήθελα να κάνω λίγα σχόλια στη βάση μιας πρώτης αξιολόγησης των πληροφοριών που λάβαμε. Πρώτα, φαίνεται ότι τα σχεδιαζόμενα έργα φαίνεται ότι εμπίπτουν στο παράρτημα 2 της οδηγίας για την μελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Τα σχεδιαζόμενα έργα τα οποία εμπίπτουν στο παράρτημα αυτό απαιτούν μόνο screening, παρακολούθηση, όχι πλήρη διαδικασία που προβλέπεται από την οδηγία. Επιπλέον, η διαβούλευση με το κοινό, η δημόσια διαβούλευση δεν απαιτείται. Επιπροσθέτως θα ήθελα να ρωτήσω τους αναφερομένους αν είναι δυνατόν να φωτίσουν δύο πτυχές. Πρώτον, δεν είναι σαφές για μας εάν η έγκριση, η άδεια δηλαδή για την ε, κατασκευή έχει ήδη δοθεί. Δεύτερο, θα είναι χρήσιμο να διασαφηθεί ποια μέσα προσφυγών έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί ενώπιον των ε, αρμοδίων εθνικών αρχών. Ευχαριστώ. Τώρα το λόγο μπορούν να λάβουν τα μέλη της Επιτροπής Αναφορών και πρώτα η κυρία Εύη. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω τους ε, αναφέροντες αυτής της αναφοράς. Είναι πολύ σημαντικό γιατί φέρνει εδώ στις Βρυξέλλες, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μια ιστορική μάχη, ένα ιστορικό αγώνα για τους πολίτες ε, του Μιλάνου και την πόλη του Μιλάνου. Γιατί το Μιλάνο είναι μια πόλη που υποφέρει από μια ποιότητα ε, πολύ κακή του ατμοσφαιρικού αέρα και επομένως εδώ και χρόνια έχει ανοίξει διαδικασία επιπερβάσεις για τα δεξίδια. Ε, του αζότου και για τα μικροσωματίδια και φυσικά δεν πρέπει να βάζουμε σε κινδύνο την υγεία των πολιτών και το να σκεφτόμαστε ότι το να χτιστεί μια τέτοια περιοχή η οποία ε, με το χρόνο η φύση έκανε τη δική της δουλειά και ε, ξανάφερε στο χώρο προστατευμένα είδη αμφιβείων και πουλιών και αποτελεί ένα πραγματικό πράσινο πνεύμονα για την πόλη μου φαίνεται μια ε, επιλογή που ε, είναι ιδιαίτερα μειοπική. Δεν κοιτάζει προς τα μπρος. Εγώ συμφωνώ με όσα υποστηρίζουν ε, οι αναφέροντες και υπογράφονται στην αίτηση. Έχουμε ένα πράσινο χώρο που πρέπει να προστατευτεί γιατί αποτελεί κοινό αγαθό και εγγυάται καλύτερο ατμοσφαιρικό αέρα, αλλά εγγυάται και ένα από τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη βιοπικιλότητα δυστυχώς ε, βλέπουμε να είναι σε κίνδυνο. Έτσι λοιπόν ε, πρέπει να τα προστατεύσουμε όλα αυτά, να προστατευτεί μια τέτοια περιοχή. Ακόμη και χρησιμοποιώντας ε, κάποιους συνδέσμους που έχουν να κάνουν με το τοπίο. Δηλαδή έχουμε και ιστορική σημασία αυτής της περιοχής. Η πιάτσα Ντάρμι νομίζω ότι θα πρέπει να ενταχθεί σε σχέδια χωροτοξικού συνδυασμού και θα πρέπει να ε, ενταχθεί ε, σε μια νομοθεσία που να αφορά και την προστασία του τοπίου για να αποφύγουμε την τσιμεντοποίηση. Πιστεύω ότι η περιοχή αυτή θα πρέπει να παραμείνει ένας δημόσιος πράσινος χώρος ε, που να προστατεύει το πράσινο και, το, και τη βιοπικιλότητα και είναι ένας από τους χώρους που θα πρέπει να ανακτηθούν διατηρώντας και την τον ιστορικό χαρακτήρα του χώρου. Να χρησιμοποιείται λοιπόν και για κοινωνικούς σκοπούς ε, η περιοχή αυτή. Δεν ε, κατανοώ ακριβώς ε, αυτά που μας είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν μας ε, έχει δώσει απαντήσεις από το Μάιο του 2018. Έχουν περάσει πολλοί μήνες και έρχεται σήμερα με μια πολύ περιορισμένη απάντηση που με εκπλήσει και μάλιστα αναφέρεται και στην οδηγία και μας λένε ότι τα έργα θα πρέπει να, να υποβληθούν απλώς σε ένα screening. Εγώ όμως ε, θέλω να πω ότι για την ε, χωροταξία, βέβαια εδώ και ο Δήμαρχος έχει σημαντικό ρόλο στο να ζητήσει την άποψη των πολιτών για το τι θα γίνει με αυτή την ε, περιοχή. Κάνω κάποιες προτάσεις για το πώς να συνεχίσουμε, Πρόεδρε, και κλείνω. Θέλω να ζητήσω να μπορέσουμε συγκεκριμένα να μεταφερθούν τα αιτήματα των πολιτών στο Δήμαρχο του Μιλάνου Ελλά και στον Περιφερειάρχη της Λομβαρδίας αλλά και στα τρία Υπουργεία που είναι αρμόδια και θα πρέπει να συμμετέχουν στην προστασία του χώρου αυτού στο Υπουργείο ε, Πολιτισμού, στο Υπουργείο Οικονομίας και το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Ευχαριστώ ουσιαστικά και εσείς προτρέχετε και είπατε ακριβώ αυτά που θέλω να πω και εγώ όταν θα φτάσω στη σύνοψη. Τώρα θα πρέπει να επιστρέψω τον λόγο, αλλά για ένα λεπτό στον αναφερόμενο, να δώσει ίσω κάποια ειδική εξήγηση, γιατί έχουμε ακόμα μία ε, αναφορά σχετική με τη Βρετανική αποχώρηση, το Brexit. Άρα, πολύ σύντομα σα παρακαλώ κύριε αναφερόμενε. Αν θέλετε, αλλιώ μπορώ να προβώ εγώ στη σύνοψη. Ευχαριστώ πα, παρουσιάστηκαν έργα για την πιάτσα Ντάρμι. Υπάρχει ένα σχέδιο που προβλέπει 290 ε, τετραγωνικά μέτρα ε, οικοδομήσιμης περιοχής. Υπάρχουν 50 ε, κτίρια με 11 κτίρια που θα ακυρώσουν για πάντα θα σκοτώσουν για πάντα μία περιοχή που είναι θησαυρό ε, βιοπικιλότητας, 5 χιλιόμετρα από το κέντρο του Μιλάνου, από την πιάτσα ε, την Τουόμο. Είναι σημαντικό και για την ε, Ευρώπη την ίδια, δεδομένου της ε, σημασίας της Μητροπολιτικής περιοχής του Μιλάνου. Γι' αυτό ακριβώς ήρθαμε εδώ, γι' αυτό γράψαμε την αναφορά. Εμείς στείλαμε στην κοινότητα του Μιλάνου πολλά έγγραφα από εμπειρογνώμονες ε, βοτανικής, ε, υδρολογίας, ε, που δείχνουν ακριβώς αυτά που ισχυριζόμαστε, αλλά δεν μας άκουσαν. Αυτά. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ για τις παρεμβάσεις σας. Θα προσπαθήσω να κάνω μια σύνοψη. Βεβαίως θα κρατήσουμε ανοιχτή την αναφορά θα αποστείλουμε επιστολές στις αρμόδιες αρχές, τα Υπουργεία όπως είπαμε πριν, διότι α, υπάρχει και νέα κυβέρνηση τώρα ε, με νέους υπουργούς οι οποίοι ε, οφείλουν να μελετήσουν το θέμα. Αναμένουμε τις ε, γραπτές απαντήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που μας υποσχέθηκε τις διαβιβάσει σύντομα και θα στείλουμε επιστολή και στο Μιλάνο, στην περιφέρεια της Λομβαρδίας και στα αρμόδια Υπουργεία σας. Αυτό μπορούμε να κάνουμε για να φωτίσουμε τα θέματα. Βλέπω ότι συμφωνεί και ο αναφερόμενος. Με το καλό να επιστρέψετε στην πατρίδα σας και σας ευχαριστούμε που ήλθατε και σας ευχόμαστε και ε, καλή επιτυχία στην προσπάθειά σας να διαφυλάξετε αυτή την όμορφη γωνιά της Ευρώπης. Τώρα το 10 που είναι η συνέχεια που δίνεται σε αναφορές πολιτών σχετικά με το Brexit. Έχουμε λάβει σχετικές αναφορές, έχουμε κάνει και ακροάσεις μαζί με την Επιτροπή Θεμελιωδών Ελευθεριών, έχουμε παρέμβει και με ψηφίσματα. Εγώ ίδια προσωπικά έχω συνεργαστεί και είμαι σε στενή επαφή με τον διαπραγματευτή για το Brexit, τον κύριο Μπαρνιέ, ως ε, συμμετέχουσα στους, ε, στην διάσκεψη των Προέδρων των ε, Επιτροπών. Έχουμε λοιπόν κάνει μεγάλη προσπάθεια για να λάβουμε υπόψη όλα τα θέματα που απασχολούν τους ε, Βρετανούς πολίτες και τους Ευρωπαίους πολίτες. Τα πάντα θα μείνουν ανοιχτά. Καμία αναφορά για το Brexit δεν πρόκειται να κλείσει. Τις κρατούμε ανοιχτές και παρακολουθούμε προσεκτικά και καθημερινά τις εξελίξεις μετά την απόρριψη δηλαδή από την Βρετανική Βουλή της ε, συμφωνίας και βέβαια και ε, την ε, επιβίωση της Βρετανικής κυβέρνησης της ψήφου της ψηφοφορίας για την πρόταση Μομφής. Θα δώσω τώρα το λόγο στην αναφερομένη, αλλά αν μπορείτε να κρατηθείτε μέσα στο όριο των τριών λεπτών, γιατί αποχωρούν οι διερμηνείς μας στις 30 ακριβώς. Παρακαλώ να είστε το δυνατόν συντομότεροι για να προλάβετε να ακούσετε και τους, άλλους, ε, και τους ευρωβουλευτές μάλλον, καθώς και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα κάνω ό,τι μπορώ. Τέσσερα λεπτά. 1,2 εκατομμύρια Βρετανοί στο όνομά τους που ζουν στην Ευρώπη. Ε, στο όνομά του σας ευχαριστώ, ευχαριστώ που μα επιτρέπετε να αναφερθούμε στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων και η Τερέζα Μέη και ο Μισελ Μπανιέ μας υποσχέθηκαν ότι τα 5 εκατομμύρια προσώπων που έχουν ασκήσει το δικαίωμά τους για μετακίνηση από τι δύο πλευρέ θα, θα βρεθούν στο επίκεντρο των προσπάθειών του. Έκτοτε όμω έχουμε μεγάλη αβεβαιότητα στο Westminster και δεν βλέπουμε να υλοποιούνται οι υποσχέσει. Πρόκειται για σημείο καμπή για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι πολίτε θεώρησαν ότι είναι αξιόπιστε οι δεσμεύσει και οι υποσχέσει για την τήρηση των δικαιωμάτων του μετά το Brexit. Η μεταχείριση που θα υποστούμε τώρα θα είναι και το μήνυμα για το μέλλον. Για το πώ δηλαδή συμπεριφέρεται η Ευρωπαϊκή Ένωση στους πολίτε τη. Πού βρισκόμαστε. Έχει αποσυρθεί η συμφωνία, μάλλον έχει κατατεθεί η συμφωνία με ειδικό κεφάλαιο για τα δικαιώματα των πολιτών που επιτρέπει για παράδειγμα στους Βρετανούς ε, πολίτες που διαβιούν στις 27 χώρες μέλη της Ένωσης να ε, συνεχίσουν να ασκούν την ε, ελευθερία του κυκλοφορήν. Αυτό είναι ουσιαστικό. Όμως η συμφωνία φαίνεται πως δεν γίνεται δεκτή από την πλευρά του Λονδίνου και σε ό,τι το αφορά είναι νεκρή. Αυτό όμως θα είναι καταστροφή για τους, Ευρω... για τους Βρετανούς στην Ευρώπη. Θα χρειαστεί να αντιμετωπίσουμε, δηλαδή εμείς οι Βρετανοί που ζούμε στην Ευρώπη, 27 διαφορετικές δικαιοδοσίες. Βρισκόμαστε μόλις λίγες εβδομάδες πριν από την ημερομηνία της Βρετανικής αποχώρησης και ακόμα δεν υπάρχουν λεπτομέρειες για την προστασία των δικαιωμάτων μας. Εξ όσου γνωρίζουμε, καμιά χώρα δεν έχει ακόμα ψηφίσει νομοθεσία που θα μας επιτρέψει να είμαστε νομίμως διαμένοντες μετά από το τέλος Μαρτίου 2019. Αναμένουμε να δούμε τώρα τις λεπτομέρειες, αλλά αυτά που ακούμε δεν μας ικανοποιούν. Από τις δηλώσεις που έχουμε ακούσει ως τώρα, κάθε χώρα μέλος θα μας αντιμετωπίσει διαφορετικά. Ορισμένες χώρες θα ε, αντιμετωπίσουν τους Βρετανούς πολίτες ως ε, πολίτες τρίτων χωρών, άλλες διαφορετικά. Σε ορισμένες ε, προτείνονται κάποιες ε, Προθεσμία έω τριών μηνών. Οι Βρετανοί πολίτε που διαμβαίνουν σε τρίτες χώρες θα διατηρήσουν για κάποιο δικαίωμα κάποια δικαιώματά του, άλλοι ίσως όχι. Εν πάση περιπτώσει πρόκειται για πλήρη σύγχυση. Θα οδηγήσει σε διαφορετικές και διακριτικέ μεταχειρήσει. και επάνω από όλα αυτά έρχεται και το ρεφρέν ότι τα δικαιώματά μας θα εξαρτηθούν από το πώ θα αντιμετωπίσει το Ενωμένο Βασίλειο τα 3 εκατομμύρια Ευρωπαίων που διαμένουν εκεί. Δεν το καταλαβαίνουμε εμείς αυτό το πράγμα. Η προσέγγιση αυτή δεν μα γεμίζει αυτοπεποίθηση. Θα υπάρξουν τεράστιες δυσχέρειες για τους Βρετανούς πολίτες που διαβιούν στις 27 χώρες μέλη. Είμαστε ένας πληθυσμός κινητικός. Εργαζόμαστε και σε πλείονες χώρες μέλη. Εάν δεν υπάρχει μια ενιαία ε, στάση των χωρών αυτών, θα έχουμε πάρα πολύ σημαντικά προβλήματα σε κοινωνικά δικαιώματα, σε συνταξιοδοτικά δικαιώματα και ούτω καθεξής, όπου έχουμε καταβάλει καλή την πίστη και τις κρατήσεις μας και ούτω καθεξής. Έχουμε λοιπόν ένα βέβαιο μέλλον και εντελώς αβέβαιο συνταξιοδοτικό μέλλον. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τα παιδιά μας, τα οποία και αυτά είναι Βρετανοί πολίτες που διαβιούν και μεγαλώνουν σε 27 ευρωπαϊκές χώρες μέλη και τους τραβάνε ξαφνικά το χαλί κατά από τα πόδια, χωρίζοντα οικογένειε. Καμιά φορά έχει δικαιώματα ένα παιδί και όχι ένα άλλο. Τι διδάσκει αυτό στην επόμενη γενιά ψηφοφόρων. Σε τέσσερι μήνες από τώρα θα αρχίσουν και οι προεκλογέ. Θα πάτε τότε στους ε, ψηφοφόρου και θα τους ε, ζητήσετε την εμπιστοσύνη τους. Ε, πώ θα σας τη δώσουν. Δεν υπάρχουν πιο ένθερμοι υποστηρικτέ τη προσπάθεια αυτή από τους Βρετανούς πολίτες που διαβιούν στις 27 χώρε μέλη. Έχουμε ασκήσει το δικαίωμα μας της ελευθερίας κυκλοφορία και έχουμε πληρώσει το τίμημα. 60 και πάνω το 100 από εμά έχουμε χάσει τα δικαιώματά μας, τα εκλογικά μας δικαιώματα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πολλοί από εμά δεν θα μπορέσουμε να επιστρέψουμε στην πατρίδα μα, Ποτέ δεν θεωρήσαμε ότι είμαστε πολίτε του πουθενά ήμασταν πολύ ε, άνετα, αισθανόμασταν πολύ άνετα στην διπλή μας ιδιότητα Βρετανών πολιτών και Ευρωπαίων πολιτών, αλλά τώρα μας απογοητεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι ε, Βρετανοί που βρίσκονται λοιπόν στην Ευρώπη θα θέλαμε να ζητήσουμε. Εάν δεν υπάρξει συμφωνία τελικά, πάρτε το τμήμα εκείνο της συμφωνίας που αναφέρεται στα δικαιώματα των Βρετανών πολιτών και περιφρουίστε το, περιφράξτε το και χρησιμοποιήστε, εφαρμόστε το αυτό, διότι αν δεν μπορούμε να ε, βασιστούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πού μπορούμε να βασιστούμε. Και αν δεν μπορούμε να βασιστούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα, πότε θα μπορούμε. Αυτή είναι και η στιγμή που καλείστε εσεί να αποδείξετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση των πολιτών. Χρησιμοποιήστε, δράξτε αυτή την ευκαιρία πριν αποδειχτεί ότι είναι πολύ αργά. Σα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρο, σα ευχαριστώ για την μεγάλη προσπάθεια και τον χρόνο που έχετε αφιερώσει στην ε, υπόθεση αυτή. Πολύ ε, αισθανόμαστε πάρα πολύ μεγάλη συμπάθεια για σας και για την υπόθεσή σας. Έχω ζητήσει και... Ε, μάλλον έχουμε προσκαλέσει και την Μόνη Κόγγενς. Σας παρακαλώ μην επαναλάβετε ωστόσο τι είπε η σα, έτσι ώστε να προλάβουμε να ολοκληρώσουμε στις 6.30 γιατί μετά δεν θα έχουμε και διερμηνία. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο εκ μέρους των ε, τριών εκατομμυρίων. Πριν ε, δύο χρόνια, πριν μια εβδομάδα, πριν να δημιουργηθεί αυτή η αναφορά, ήμουν ε, μέρος μιας αντιπροσωπείας των τριών εκατομμυρίων που κλήθηκαν να συναντηθούν με τον κύριο Μπαρνιέ στη συνεδρίαση. Μας εξήγησε ότι τίποτα δεν έχει συμφωνηθεί μέχρι να συμφωνηθούν όλα και με ένα τεράστιο σοκ από ό,τι κατάλαβα μας χρησιμοποιούσε σε ένα διαπραγματευτικό χαρτί και ε, τώρα ε, μας παρουσιάζουν ένα του Ηνωμένου Βασιλείου αν ε, δεν συμφωνήσει να εφαρμόσει τη Συμφωνία Αποχώρησης και εδώ σκέφτομαι, παραδείγματος χάρη, κάποια δικαιώματα ελεύθερης μετακίνησης. Ε, δυστυχώς, εμείς θεωρούσαμε ότι θα πρέπει να προστατευμένα τα δικαιώματά μας. Τι εννοούμε με την προστασία αυτή, η Rick Fencing. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να συμφωνήσουν η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Μένο Βασίλειο να δεσμευτούν στο να εφαρμόσουν το μέρος της συμφωνίας ε, που αφορά τα δικαιώματα των πολιτών, ε, όπως και να έχει, ακόμη και δεν υπάρχει συμφωνία σε άλλες πτυχές. Ε, μόνο έτσι θα προστατευτούν τα δικαιώματα όλων μας από την ε, διεθνή συνθήκη παρά από την εσωτερική εθνική νομοθεσία και για τα 3 εκατομμύρια που δεν θα έχουν προστασία από τέτοιες διεθνείς συμφωνίες, οι συνέπειες θα είναι δραματικές. Και εδώ δημοσιεύτηκε από το Ηνωμένο Βασίλειο ένα έγγραφο πολιτικής για το τι θα γίνει με τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αν δεν υπάρχει ε, συμφωνία. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει συμφωνία, λέει ότι δεν μπορούμε να ζητήσουμε θα γίνει ενώ, παραδείγματος χάρη, εγώ έχω διασφαλίσει ε, το δικαίωμά μου αν η μητέρα μου μπορεί να έρθει στο Ηνωμένο Βασίλειο από την Ολλανδία αν με χρειαστεί και λέει το Ηνωμένο Βασίλειο όχι. Δημοσιεύτηκε και μια νομοθεσία νομοθεσία για τη μετανάστευση και ε, θέλει ουσιαστικά να εξαλείψει από τη Βρετανική νομοθεσία κάθε ίχνος ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την ελεύθερη μετακίνηση. Ε, τα δικά μας δικαιώματα θα αναφέρονται σε μεταναστευτικούς κανόνες. Θα είναι δευτερογενική νομοθεσία που θα προσαρτώνται σε κοινοβουλευτική πράξη και θα μπορούν να αλλάξουν οι κανόνες αυτές χωρίς κανένα κοινοβουλευτικό έλεγχο. Μεταξύ του 2012 και τώρα αυτοί οι κανόνες άλλαξαν 65 φορές οι αλλαγές αυτές δημοσιεύτηκαν απλώς κάπου και αν ε, κάποιος ε, στο κοινοβούλιο ε, δεν έφερε αντίρρηση έγιναν νόμος. Έτσι λοιπόν αυτό οδηγεί σε δυνατότητες σύλληψης και απέλεσης πολλών πολιτών χρειάζεται, χρειάζονται οι Ευρωπαίοι πολίτες ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο ε, προστασία διαβίου. Αν τρία εκατομμύρια πολίτες ε, αφαιθούν στο τι αποφασίσει το κράτος αυτό και όλα τα δικαιώματά τους μπορούν να αφαιρεθούν, τότε κουρουλιάζει την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλω να ζητήσω λοιπόν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ασκήσει όση επιρροή έχει στους 27 αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων και στο Συμβούλιο για να πράξουν το σωστό για να δώσουν εντολή στην Κομισιόν να ε, έρθει σε επαφή με το Ενωμένο Βασίλειο για να διαφυλάξει τη Συμφωνία για τα Δικαιώματα των Πολιτών και να δεσμευτεί να την εφαρμόσει υπό το άρθρο 50, όπω και να έχει. Ενώ και τώρα, ακόμη και αν υπάρχει παράταση του άρθρου 50 και σε σχέση με το να κάνετε το σωστό, θέλω να ασκήσετε την επιρροή σα προκειμένου να διασφαλίσετε πλήρη δικαιώματα ελεύθερη μετακίνηση ε, για του ε, Βρετανού φίλου μα. Αυτό θα πρέπει να γίνει τουλάχιστον. Thank you very much. Now I'm... Σας ευχαριστώ. Τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στον κύριο Αρμπό. Ξέρω ότι είναι πολύ λεπτό το ζήτημα. Είμαστε σε καθημερινές επαφές με τον Μισελ Μπαρνιέ για το θέμα αυτό. Επομένω, ε, εντάξει, δεν χρειάζεται να αισθάνεστε πίεση, απλώ εν συντομία να μα ενημερώσετε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και για τα καλά σα λόγια ευχαριστώ. Θα είμαι πολύ σύντομο. Θα μπορούσα να πω πάρα πολλά, αλλά δεν έχουμε και χρόνο. Ξέρουμε φυσικά τι ανησυχίε που υπάρχουν, ε, ειδικά από του πολίτε που να ασκήσουν το δικαίωμα ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, θα θέλανε αυτά τα δικαιώματα να υπάρχουν για πάντα. Παρά τις προσπάθειες που κάνουμε, οι άνθρωποι αυτοί, ε, από τη στιγμή που θα γίνει η αποχώρηση, ε, οι πολίτες αυτοί θα γίνουν υπήκοοι τρίτων χωρών, οι Ευρωπαίοι πολίτες δεδομένως, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μετριάσουμε το αποτέλεσμα της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου, ε, για 4,5 εκατομμύρια Ευρωπαίους πολίτες ε, που θα επηρεαστούν ήταν από τις πρώτες προτεραιότητες από την πρώτη μέρα και ήταν ε, στην καρδιά της εντολής που δόθηκε στις διαπραγματεύσεις. Θα πρέπει τα δικαιώματα των πολιτών να είναι προϋπόθεση για να διευρύνουμε τη συζήτηση σε άλλα θέματα. Στις 17 Σεπτεμβρίου ε, Δεκεμβρίου ε, συμφωνήσαμε επί της αρχής με το Νομένο Βασίλειο για την εξασφάλιση των πλέον σημαντικών δικαιωμάτων αυτών των πολιτών που θα πληγούν και αυτό ε, οδήγησε στο σχέδιο συμφωνίας του, που επικυρώθηκε από το Κοινοβούλιο στις 25 Νοεμβρίου. Ε, ήμασταν πάντα διαφανείς στην όλη διαδικασία και ήρθαμε σε επαφή και με τους, ε, και τις οργανώσεις και τους ε, Βρετανούς πολίτες στην Ευρώπη. Ε, με βάση τη συμφωνία αποχώρησης, εστιάσαμε στο στόχο να εγγυηθούμε σε αυτούς τους πολίτες μάλλον να ασκούν το δικαίωμα ελευθερής κυκλοφορίας, παραμένοντας και κατοικώντας εκεί, και κρατώντας ε, το δικαίωμά τους αυτό μέχρι την καταληκτική ημερομηνία. Ε, Διαφυλάσσει τα δικαιώματα των ε, κατοίκων, τα δικαιώματά τους ως αυτοαποσχολούμενων και εργαζόμενων, καθώς και το δικαίωμα ίσης μεταχείρισης, καθώς και συντονισμό για θέματα κοινωνικών ασφαλίσεων. Για την αποτελεσματικότητα αυτών των δικαιωμάτων τώρα. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες. Υπάρχουν διάφορες διατάξεις στη Συμφωνία Αποχώρησης που θα εξασφαλίσει ότι αυτά τα δικαιώματα θα είναι εφαρμοστέα και μπορεί να τα ασκήσει κανείς. Φυσικά υπάρχει μια βεβαιότητα, την ξέρουμε όλοι, την αναφέρατε κι εσείς, ε, για το ring fencing. Ήταν ο βασικό στόχο του Μπαγνιέ να εξασφαλίσει τα δικαιώματα των πολιτών. Ακούμε βεβαίως ότι θα πρέπει ίσως ε, γύρω από τα δικαιώματα των πολιτών να καταλήξουμε σε μια μήνυ συμφωνία, ούτω ώστε να διαφυλάξουμε αυτά τα δικαιώματα. Ε, εμείς πιστεύουμε ότι θα ήταν λάθος αυτό, ότι ο καλύτερος τρόπος για να προστατεύσουμε 4,5 εκατομμύρια πολίτες είναι να βρούμε μια συνολική συμφωνία. Ο καλύτερος τρόπο για να το πετύχουμε αυτό δεν είναι κατά την απόψή μα να αποδεχτούμε την αποτυχία των διαπραγματεύσεων που θα σήμαινε ότι παίρνουμε μια νέα κατεύθυνση και πάμε προς το ring fencing, γιατί ring fencing σημαίνει παραδοχή της αποτυχίας. Ε, σε περίπτωση ε, μη συμφωνίας, το Ηνωμένο Βασιλείο είπε ότι τα βασικά δικαιώματα των ε, ατόμων αυτών θα διασφαλιστούν στο Ηνωμένο Βασίλειο, δηλαδή θα πρέπει να δούμε τις λεπτομέρειες. Σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Κομισιόν είπε το Νοέμβριο, 30 Νοεμβρίου, και αρχές ε, Δεκεμβρίου ότι θέλει μια ε, γενική συμφωνία των κρατών μελών σε περίπτωση no deal. Όμως ε, μπορεί σε περίπτωση που δεν υπάρχει συμφωνία ο καθένας να προβεί σε μονομερείς ενέργειες. Αλλά και τα δύο μέρη είπαν ότι σε αυτήν την περίπτωση θα προστατεύσουν τους ανθρώπους, απλώς δεν ξέρουμε περισσότερες λεπτομέρειες σε αυτή τη φάση, γιατί εστιάζουμε ακόμα τις προσπάθειές μας ε, στο σενάριο της διαπραγμάτευσης. Δεν, θέλω να, δεν θέλουμε ακόμα να παραδεχτούμε ότι δεν υπάρχει συμφωνία, ότι υπάρχει no deal. Γιατί αυτό ε, νομίζω ότι υποσκάπτει την πιθανότητα έφτακτης αποχώρησης, ε, συντεταγμένης αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου. Now the floor is open to, to, um, to... Τώρα να δώσουμε το λόγο στους συναδέλφους. Πρώτα η κυρία ε, Κέρτον Πρώτα θα ήθελα να αποτίσω φόρο τιμή στα 3 εκατομμύρια Βρετανών για την αξιοπρεπή εκστρατεία που ζουν εδώ στην Ευρώπη δηλαδή, που έκαναν τα τελευταία χρόνια στα πλαίσια αυτά μεγάλου άγχους και αβεβαιότητας που καθιστά πολύ δύσκολο για πολλούς να κρατήσουν την ψυχραιμία τους και δυστυχώς πολλοί στην Βρετανία δεν αντιλαμβάνονται την ψυχολογική επίπτωση Τη απόφασης που λάβαμε το 2016 ως χώρα, εννοεί το δημοψήφισμα, τις επιπτώσεις ε, στην ζωή των ανθρώπων, στην ε, ψυχολογική και ε, διανοητική του υγεία. Από τι λοιπόν φόρο τιμή και στις δύο οργανώσεις, άνθρωποι οι οποίοι συνέρχονται εθελοντικά για να βρουν λύσεις. Τρέχει ο χρόνο και, και σήμερα εδώ τρέχει και ο χρόνο για το Brexit. Και μένει λίγο χρόνο πριν από τι 29 Τρίτου, ώστε να προλάβουμε να τα κάνουμε όλα αυτά τα πράγματα και γι' αυτό. Και ιδίω έχοντα ακούσει την Πρωθυπουργό μα στην Βουλή των Κοινοτήτων σήμερα το απόγευμα να λέει ότι το εναλλακτικό σχέδιο στην πραγματικότητα είναι το πρώτο σχέδιο, δηλαδή δεν υπάρχει plan B και δεν υπάρχει καμία απολύτω αλλαγή στι προτάσει τη, παρόλη την ιστορική τη ήττα στην Βουλή των Κοινοτήτων, η Ευρώπη των 27 Φοβούμαι ότι θα πρέπει να φανεί ότι είναι ο ενήλικος μέσα στο δωμάτιο, ας το πω έτσι. Μαζί με ένα μεγάλο αριθμό των συναδέλφων μου, Βρετανών Ευρωβουλευτών από διάφορα κόμματα, συντάξαμε επιστολή στον πρόεδρο Τούσκ, στον κύριο Μπαρνιέ, στον πρόεδρο Ιούνκερ και στον κύριο Βερχόφστατ, ζητώντας κατά βάση από την Ευρώπη των 27 να δώσει μονομερός εγγύηση στους Βρετανούς πολίτες που διαβιούν στην Ευρώπη για τα δικαιώματά τους, έτσι ώστε να αναγκάσει την, Ευρω... την Βρετανική κυβέρνηση να πράξει το ίδιο για τους Ευρωπαίους που διαβιούν στο Ηνωμένο Βασίλειο. το κόστος ε, της ε, ε, ρύθμισης του καθεστώτος των προσώπων αυτών είναι πολύ λιγότερο από το κόστος του Brexit. Είναι πολύ περιορισμένος ο χρόνος που έχουμε στη διάθεσή μας για να ρυθμίσουμε τα πράγματα. Φοβούμε ότι η χώρα μου και η κυβέρνησή της δεν είναι αρκετά όρημη και ενήλικη ώστε να παίξουν σωστά το ρόλο. Απευθύνω λοιπόν έκκληση στους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ηγούνται των διαπραγματεύσεων να δείξουν υπεύθυνη στάση και να βάλουν σε πρώτη θέση τα δικαιώματα των πολιτών, διότι έτσι θα δείξουν την αξία του ευρωπαϊκού ε, ε, σχεδίου ολοκλήρωσης. Αν δεν μπορούμε να υπερασπιστούμε τα δικαιώματα των πολιτών μας, τότε πραγματικά βρισκόμαστε σε πολύ άσχημη κατάσταση. Σας ευχαριστώ, Τζουντ. Η κυρία Μούντι. Ευχαριστώ πολύ. Μάλλον θα ακούσετε τα ίδια σχόλια, αλλά όπω ε, και Τζούτι, θα ήθελα να ευχαριστήσω του αναφέροντε για την εξαιρετική εκστρατεία και ευχαριστώ και εσά, Πρόεδρε, γιατί ξέρω ότι στο ρόλο σα ω Πρόεδρο στην ε, συνεδρίαση των Πρόεδρων των Επιτροπών ε, έχετε υποστηρίξει αυτό το ζήτημα συνεχώς. Ως εκπρόσωποι στον Ομένο Βασίλειο λαμβάνουμε συνεχώς επιστολές από ανθρώπους που ζουν ε, τώρα σε άλλες χώρες αλλά και από Ευρωπαίους που ζουν στις ε, δικές μας εκλογικές ε, περιφέρειες και πραγματικά κάποιες ιστορίες είναι ιδιαίτερα συγκινητικές και είναι τρομερές οι εμπειρίες που είχαν οι άνθρωποι ως συνέπεια του τι συμβαίνει στο Ηνωμένο Βασίλειο. συνέπειε του δημοψηφίσματο, δηλαδή. Είναι σημαντικό όλοι ε, να είμαστε εδώ και να υποστηρίζουμε αυτούς τους ανθρώπους και να αποτελούμε τη φωνή των ανθρώπων αυτών, οι οποίοι βιώνουν κάτι που δεν θέλουν καθόλου να συμβεί, αλλά ε, δυστυχώς τους επιβάλλεται. Και καθώς ε, σήμερα το απόγευμα συζητάμε εδώ και έχουμε όλα τα συμβαίνουν στο Westminster με το σχέδιο Α να γίνεται σχέδιο Β και πάλι σχέδιο Α και δεν ε, υπάρχει καμία απτή αλλαγή μετά από αυτή την ιστορική ήττα. Είναι απαραίτητο τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει το σωστό για τους ε, Ευρωπαίους πολίτες και για τους πολίτες που πιστεύουν στην ιδέα της Ευρώπης. Έτσι λοιπόν ε, πηχώ όσα υπόθηκαν από τις αναφέρουσες αλλά και από την Τζουντ. Τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να δείξει το θάρρος της ε, και την πεποίθησή της ε, και να δεσμευτεί απέναντι σε αυτούς τους πολίτες προκειμένου να γίνουν σεβαστά πλήρως τα δικαιώματά τους. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε ακόμη τέσσερα λεπτά από τους διερμηνείς. Σας ευχαριστώ πολύ. Μετά από αυτό, αν θέλετε, μπορείτε να αποχωρήσετε, γιατί εμείς ούτως ή άλλως ε, μιλάμε και αγγλικά στην αίθουσα. Εγώ προσωπικά θα ήθελα να συνεχίσουμε για να καταγράψουμε και τις δηλώσεις. Παρακαλώ. Ε, κυρία Σκοτ κάτω. Ευχαριστώ. Θα είμαι σύντομη για να μην ε, ξοδέψω πολύ από το χρόνο σας. Θα ήθελα και εγώ να συμφωνήσω. Έχετε κάνει εξαιρετική δουλειά ε, στην εκστρατεία σας ε, και συμφωνώ ότι με βγαίνει τρόπο έχετε τη δράση ενώ σας έχουν οθήσει σε μια τρομερή κατάσταση πέραν ελέγχου. Θα ήθελα να αμφισβητήσω κάτι που εκπρόθηκε από την Κομισιόν. Δεν εκπροσωπείται εδώ τον κύριο Μπερνιέ, αλλά θα ήθελα αυτό να το αναφέρετε, γιατί εδώ έχουμε μια κατάσταση που έχουμε εμ, ανάγκες ε, και ωφέλη και στις δύο πλευρές, ισότιμες, αντίστοιχες, ε, για δύο ομάδες πολιτών. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει τίποτα που θα χαθεί ή που θα κερδιθεί αν μπορέσουμε να αντιστοιχίσουμε τις ανάγκες αυτών των πολιτών και συμφωνήσουμε για τους πολίτες που παραμένουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν ε, βλέπω κάποιο λόγο να μην το κάνουμε και αν ε, ο λόγος ε, είναι απλώς να ασκήσουμε πίεση, τότε δυστυχώς δεν μπορούμε να κρατάμε ομοίρους τους πολίτες. Είναι εξοργιστικό. Έτσι λοιπόν, νομίζω ότι οι άνθρωποι θα πρέπει να τη χάνουν διαφορετικές μεταχείρισεις, θα πρέπει να έχουν γίνει να έχουν γίνει σεβαστά και να προστατεύονται τα δικαιώματά τους ε, γιατί ε, μιλάμε και για τους ε, ε, Βρετανούς πολίτες που μένουν τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους ε, Ευρωπαίους πολίτες που διαμένουν τώρα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Ward. Χαίρομαι που κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Εγώ δεν είμαι εδώ στην Επιτροπή. Πάρα πολλοί έρχονται και καταθέτουν μαρτυρίες από τις ε, τρομερές ε, εμπειρίες ε, που έχουν βιώσει, το άγχος τους και πολλές φορές έρχονται εδώ να παρουσιάσουν και λύσεις. Και δεν είναι αβοήθητα θύματα οι άνθρωποι, αλλά έρχονται και μας παρουσιάζουν λύσεις. Η ιδέα μονομερών εγγύσεων που θα μπορούσε να δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα σημαντικό στοιχείο εγώ μάλιστα ε, έθεσα και ένα γραπτό ερώτημα στον Ντόναλτ Τούσκ γι' αυτό. Το 2017 ε, δεν ε, είχε συμφωνήσει, αλλά πρόκειται για ένα θέμα που συζητεί το πολύ καιρό. Επομένως, τώρα δεν παρουσιάζουμε απαραίτητα κάτι καινούριο, παρουσιάζουμε κάτι που ήδη έχει τεθεί σε υψηλότατο επίπεδο. Έτσι λοιπόν ότι είναι σημαντικό αυτή, είναι σημαντική αυτή η επιστολή, όμως είναι πίεση παρόμοια που ήδη έχει ασκηθεί στους ανθρώπους ε, τα τελευταία δύο χρόνια. Εγώ, από τη δική μου πτυχή, θέλω να πω το εξής. Αν υπάρχει κάποιος που θεωρεί ότι δεν προστατεύονται τα δικαιώματά του μέσω των διαδικασιών που λαμβάνουν ε, τώρα χώρα, ε, τότε είναι ένας ακόμα. Και στη Συμφωνία του Δεκεμβρίου έμαθα ότι τα υιοθετημένα παιδιά δεν θα προστατεύονται από το κείμενο που είχε ε, υποβληθεί σε εμάς για να ψηφίσουμε. Και πραγματικά δεν αισθάνθηκα καλά με αυτό. Και τι εννοώ ότι οι συγκεκριμένες ε, περιστάσεις και ιδιαιτερότητες ε, των οικογενειών καλύπτουν τόσο μεγάλο φάσμα και δεν μπορούμε καν να φανταστούμε πόσο πολύπλοκη μπορεί να είναι η οικογενειακή ζωή. Ακόμη και αν τα δικαιώματα ενός ε, πολίτη δεν προστατεύονται, για μένα οπωσδήποτε πρέπει να κάνουμε κάτι έτσι ώστε να διασφαλίσουμε ότι κανένας δεν βρίσκεται σε βάλωτη κατάσταση και δεν, γίνονται, και δεν προστατεύονται τα δικαιώματά του.